Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στο σημείο 5 της ημερήσιας ε, διάταξης και πάλι ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Γκουλτιέρη, του πρόεδρου μας που δεν μπορεί να είναι εδώ, οπότε αναλαμβάνω εγώ να προεδρεύσω αυτής της τόσο σημαντικής συνεδρίασης. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που μπορώ να καλωσορίσω εδώ την κυρία Κριστίν Λαγκάρτ που είναι υποψήφια για τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως γνωρίζουμε, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Επιτροπής, ο τωρινός ο κύριος Δράγκη, αποχωρεί την 21 η Οκτωβρίου μετά από πέντε χρόνια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 283 σημείο 2 της ε, Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί μετά από σύσταση του Συμβουλίου για τον ορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα έχουμε αυτήν την ε, δημόσιο ακρόαση. Προηγουμένως ε, υποβλήθηκαν γραπτά κάπου 76 ερωτήσεις και θα βρείτε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις της κυρίας Λαγκάρτα στο σφακέλου σας. Στις 6 θα ψηφίσουμε σήμερα και μετά θα υποβάλουμε πρόταση προς απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου για τον ορισμό της κυρίας Λαγκάρτα στη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και στην σύνοδό του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 16 με 19 Σεπτεμβρίου θα ε, ψηφίσει επ' αυτού. Θα ακούσουμε για 10 λεπτά την κυρία Λαγκάρτ και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο ευρωβουλευτών που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις, οπότε εγώ θέλω να προσπαθήσω να προλάβουμε να έχουμε και λίγο χρόνο για το catch the στο τέλος. Οπότε ζητώ στην κυρία Λαγκάρτ να τηρήσει το χρόνο της, όπως και εσείς βέβαια, και να είσαστε ρεαλιστές. Αν πιστεύετε ότι με την ερώτησή σας μπορείτε να έχετε και κάποιες ουσιώδεις απαντήσεις, κάντε την. Λοιπόν, 10 λεπτά καταρχήν η κυρία Λαγκάρτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα αρχίσω ε, ζητώντα ε, κάποια πίκη από εσά. Γιατί εγώ είχα ετοιμάσει 15 λεπτά παρέμβαση. Το συζήτησα χθε με τον κύριο Γκουαλτιέρη και νόμιζα ότι είχα 15 λεπτά στη διάθεσή μου. Αλλά αν πρέπει να σταματήσω στα 10, θα σταματήσω στα 10. Κανένα πρόβλημα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ στην ε, Επιτροπή σας. Και ομολογώ ότι αισθάνομαι και κάπως ε, περίεργα συναισθαλμένα εδώ, γιατί Πολλοί από εσά έχουν βρεθεί κάποια φορά στην δικιά μου θέση, δηλαδή είσαστε υποψήφοι για κάποια θέση, σιγά σιγά μαθαίνετε και σιγά σιγά αποκτάτε τον ε, ενθουσιασμό που χρειάζεται για να εξυπηρετήσετε το σκοπό σας. Πιστεύω ότι οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Νομισματικής Ένωσης. Η κεντρικοί τραπεζίτε είναι ανεξάρτητοι. Δεν εκλέγονται όμως απευθεία από τον κόσμο. Οπότε λογοδοτούν μόνο σε αυτούς οι οποίοι εκλέγονται άμεσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί στον ορισμό μου. Σήμερα το πρωί δίστασα αν ήθελα να σας παρουσιάσω την ευρωπαϊκή οικονομική κατάσταση, να σας δώσω μια τεχνική κατάσταση για την νομισματική πολιτική. Και αποφάσισα ότι είναι ίσως πιο ενδιαφέρον να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην επαγγελματική μου εμπειρία και το υπόβαθρο που έχω και που σχετίζεται με τα καθήκοντά μου εφόσον αναλάβω την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήμουν λοιπόν επικεφαλής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα τελευταία 8 χρόνια και είχα το προνόμιο να είμαι επικεφαλής ενός οργάνου που βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής ασφάλειας ε, στον κόσμο και συνεργάζεται με τις κεντρικές τράπεζες. Επίσης ήμουν υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας και τότε συνέφερα στην επίλυση κρίσεων με εργαλεία, με ρυθμίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, έχω συμμετάσχει στην ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τώρα, τι είναι αυτό το οποίο με οδήγησε να αναλάβω τα καθήκοντα αυτά. Πρώτα απ' όλα ήμουνα αποφασισμένη και πίστευα και πιστεύω ακόμα ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρει κανείς στο κοινό και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου. Δυστυχώς έμαθα τις αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης ρυθμίσεων ή της έλλειψης αποφάσεων και πόσο αρνητικά επηρεάζουν το κόσμο. Και κατάλαβα ότι οι αποφάσεις των ε, θεσμών επηρεάζουν πάρα πολύ τις ζωές του κόσμου. Από τις θέσεις που κατήχα κατά το παρελθόν, πάντα πίστευα ότι οι αποφάσεις αυτές είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε και στην ε, μείωση των ανισοτήτων, ε, να προστατεύσουμε ε, το περιβάλλον από την κλιματική αλλαγή, να φροντίσουμε για μια ανάπτυξη με τη συμμετοχή όλων. Αυτά όλα μπορεί να μην θεωρούνται τα κύρια καθήκοντα που είναι μακροοικονομική πολιτική. Όμως τελικά πιστεύω ότι θεωρούνται και μακροοικονομικά στοιχεία σήμερα. Μια καλή ηγεσία δεν σημαίνει μόνο ότι θέτουμε προτεραιότητες, σημαίνει επίσης ότι ακούμε και ακούμε όλες τις ε, φωνές, όχι μόνο των εμπειρογνωμόνων, των ειδικών, αλλά όλων. Και επίσης βασιζόμαστε και στη διαφοροποίηση της σκέψης. Στο Διεθνές μεσοτικό Ταμείο συνεργάστηκα στενά με σημαντικούς οικονομολόγους, προκειμένου να μας δίνουν στοιχεία που βασίζονται σε δεδομένα και άκουσα πάντα προσωπικά και το προσωπικό, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια σύγχρονη προσέγγιση του έργου μας, προκειμένου να συμμετέχουν περισσότερο όλοι στο έργο του Διεθνούς Μασνατικού Τομείου και να βοηθήσουμε την κοινωνία. Αυτή ήταν η στρατηγική μου. Και γιατί συνεχίζει να είναι, γιατί ακριβώ αυτές οι ίδιες ε, αξίες είναι στις οποίες εξακολουθώ να πιστεύω και θα προωθήσω εφόσον τελικά επικυρωθεί η θέση μου στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να αναφερθώ σε τρεις αρχές που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές στο μελλοντικό μου έργο. Οι πρώτες ε, δύο που θα εξετάσω μαζί είναι η δέσμευση υπέρ της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζης. Η δεύτερη είναι η ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Αυτά τα δύο θα τα συζητήσω μαζί σας μαζί. Και το τρίτο είναι η συμμετοχή όλων να μην υπάρχουν αποκλεισμοί δηλαδή και θα σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Λοιπόν, δέσμευση και ευελιξία. Γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε από δεκαετία θεωρία και πράξη, ότι μια σαφή εντολή για την νομισματική πολιτική είναι πολύ βασική όπως επίσης και η δέσμευση της Κεντρικής Τράπεζας να πετύχει τους στόχου τη. Και αυτό το έχει δείξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την αρχή. Τα πρώτα χρόνια απέτυχε να ηγηθεί μιας ε, νομισματικής ένωσης με πάρα πολλές ε, διαφορές, κρατώντας ε, χαμηλά και σταθερό τον πληθωρισμό. Και μετά φτάσαμε το 2008 που έπρεπε να αντιμετωπίσει όχι τον πληθωρισμό αλλά τον αποπληθωρισμό. Και πάλι όμως η δέσμευσή της και η αποφασιστικότητά της ήταν ζωτική σημασία προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των τιμών σε μια περίοδο χαμηλού πληθωρισμού. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσαρμόστηκε στις νέες προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει. Οπότε ξεπέρασε τις παλιές πεπιθήσεις με τις νέες εμπειρίες και ήταν καινοτόμο στην πολιτική της με τη νέα της εργαλειοθήκη στα πλαίσια βέβαια πάντα που θέτει ο νόμος και η εντολή της. Και ακριβώς αυτή, αυτή η προσαρμοστικότητα, αυτή η ευελιξία που απέδειξε ότι διαθέτει βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συνθήκες. Χωρίς αυτήν τη δυνατότητα καινοτομίας και προσαρμογής, σίγουρα η κρίση, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των περισσότερων εμπειρογνωμόνων, θα ήταν πολύ χειρότερη. Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε επίσης κάποιες έρευνες για να εκτιμήσει τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε υπάρξει αυτή η καινοτομία, αν δεν είχε αντιμετωπίσει με προσαρμοστικότητα την κρίση. Ε, λοιπόν η οικονομία θα ήταν κατά 2% σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι τελικά. Αν, δίχα, αν δεν είχε ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2014 μη συμβατικά μέτρα. Ήταν πολύ σημαντικό που λήφθησαν και τέτοια μέτρα. Η απασχόληση επίσης βελτιώθηκε κατά 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης μετά από τα μέσα του 2013, γιατί ακριβώ αυτά τα μη συμβατικά μέτρα δημιούργησαν και πάλι εμπιστοσύνη στον κόσμο. Εφόσον επιβεβαιωθεί η θέση μου σε επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λοιπόν, θα ακολουθήσω αυτές τις αρχές. Την ε, δέσμευση αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για προσμαστικότητα, για ευελιξία ε, σε σχέση με τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται γύρω μας. Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε βέβαια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχουν εξαφανιστεί. Η Ευρωζώνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους που έχουν να κάνουν κυρίως με εξωτερικούς παράγοντες και ο πληθωρισμός παραμένει, εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός και σίγουρα πιο χαμηλός από τον στόχο. Συμφωνώ λοιπόν με την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι χρειάζεται μια πολιτική προσφοράς χρήματος προκειμένου ο πληθωρισμός να επιστρέψει στο περίφημο κάτω αλλά κοντά στο 2%. Όμως υπάρχουν και μερικά σημαντικά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας και που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η νομισματική πολιτική. Πρώτα απ' όλα, ότι οι επιπτώσεις των μη συμβατικών πολιτικών να εξακολουθούν να είναι θετικές και για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ε, για τις αρνητικές παρενέργειες, για τις παρενέργειες που μπορεί να προκληθούν από τέτοιες πολιτικές και να λάβουμε υπόψη μας και τις ανησυχίες του κόσμου. Παραμένουμε λοιπόν δεσμευμένοι στην εντολή μας που είναι για σταθερότητα τιμών, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση ε, κόστους και ωφέλους. Δεύτερον, το περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων επίση θέτει ερωτήματα στρατηγικής για όλε τι κεντρικές τράπεζες, όχι μόνο την ευρωπαϊκή. Οι κεντρικές τράπεζες λοιπόν πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα ποια είναι η δυναμική του πληθωρισμού και να χρησιμοποιήσουν νέα μέσα τα οποία μπορούν να περιορίσουν την κρίση και να χρησιμοποιήσουν ε, ισολογισμούς και μη συμβατικές πολιτικές. Και πρέπει επίσης να προβληματιστούν για το κατά πόσο τα δικά τους νομισματικά πλαίσια πολιτικής είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουν μελλοντικέ προκλήσεις. Και αυτό είναι ένας στόχος που εγώ θα αναλάβω εφόσον ε, αναλάβω επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τρίτον, οι κεντρικές τράπεζες όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουν νέα είδη προκλήσεων. Κλιματική αλλαγή, ε, τεχνολογικές αλλαγέ κατακαιρματισμός της πολυμερούς ε, τάξης που έχουμε σήμερα στον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό η νομισματική πολιτική να βλέπει μακριά και να λαμβάνει υπόψη της ε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να πετύχει τη σταθερότητα των τιμών, που είναι και εντολή τη. Τέλος, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής μας πολιτικής έχει να κάνει με την αντοχή του ε, χρηματοπιστωτικού συστήματος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ρόλο τη όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει ενισχυθεί. Τη ζητήθηκε να αναλάβει νέε αρμοδιότητε για μακροπροληπτική πολιτική και να ε, αναλάβει και ε, να προσκαλέσει μάλλον και να έχει κάτω από την αιγίδα τη ε, και την Ευρωπαϊκή Εποπτεία Τραπεζών, τη οποία τον επικεφαλή είχατε πριν από λίγο εδώ ενώπιον σα. Υπάρχει λοιπόν ο, η εποπτεία αυτή που είναι η νέα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας και ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει βελτιώσεις, έχουν μειωθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι περισσότερες ε, σημαντικές ε, τράπεζες έχουν μειώσει κατά το ίμιση τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που διαθέτουν. Όμως οι προκλήσεις παραμένουν και η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Κεφαλαιογορών πρέπει να ολοκληρωθούν και να υπάρχει έτσι βελτίωση όσον αφορά την πρόσβαση σε χρήμα. Υπάρχει χαμηλή κερδοφορία επίσης και το τοπίο αλλάζει συνεχώς γιατί οι μη τράπεζες απεκτούν όλο και σημαντικότερο ρόλο ως διαμεσολαβητές. Το μερίδιο των ε, μη τραπεζών σε σχέση με τις τράπεζες από 30% που ήταν πριν την κρίση σήμερα είναι 50%. Αυτές είναι τεράστιες αλλαγές που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν σκεφτόμαστε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι επιχειρήσεις δημοσιονομικής τεχνολογίας επίσης έχουν το 1 τέταρτο του κλάδου στη θέση του σήμερα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον και οι κεντρικέ τράπεζε και οι επόπτε πρέπει να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά να είναι και ανοιχτοί σε ευκαιρίε που προσφέρουν οι αλλαγέ αυτέ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση όσον αφορά του ε, κινδύνου για να αποφεύγουμε κλιματικές δραστηριότητες, να προστατεύουμε τον ιδιωτικό βίο, να διασφαλίζουμε την εφαρμογή των ε, ρυθμίσεων και να προστατεύουμε τα δημόσια καθά. Αλλά σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στα ωφέλη από τα οποία μπορεί να υποφεληθεί η κοινωνία εξαιτία καινοτομιών. Οπότε είπαμε δέσμευση, να είμαστε πιστοί στην εντολή μας, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και κάτι άλλο που βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η συμμετοχή όλων, να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Η πρώτη πτυχή του όρου αυτού κατά τη γνώμη μου είναι η συμμετοχή και η συνεργασία. Μέσα στο ευρωσύστημα υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που μπορεί να μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε μελλοντικέ προκλήσει. Ένα παράδειγμα είναι το πρασίνισμα των δημοσιονομικών. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ε, για αυτό το σκοπό το 2017 που συμμετέχουν οι κεντρικοί τραπεζίτες και επόπτες και αποτελεί μέλος του δικτύου αυτού και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν επίσης να παίξουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να ενισχύσουν την συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και να βοηθήσουν την πολυμερή τάξη σε όλου του τομεί των αρμοδιοτήτων τη. Οι κεντρικές τράπεζες δεν δρούν μέσα σε ένα κενό. Πρέπει να φροντίζουν για την ε, αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, η οποία μπορεί να ενισχυθεί εφόσον έχουμε τις κατάλληλες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και εφόσον υπάρχει η εμπιστοσύνη του κοινού. Γι' αυτό λοιπόν βλέπω πολλά περιθώρια για παρετέρω συνεργασία σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς επίσης, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, πρέπει να προχωρήσει, αλλά να διασφαλίσουμε επίσης και την προστασία των ε, καταναλωτών αποφεύγοντας το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό ισχύει τόσο στην πραγματική οικονομία όσο και στι υπηρεσίε, αλλά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα για τον οποίο μιλήσαμε πριν. Ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη. Ένα άλλο τομέα συνεργασία είναι οι δημοσιονομικέ πολιτικέ, που πρέπει να βοηθούν τη σταθεροποίηση των οικονομιών μα και να αποφεύγουν τον υπερβολικό φόρτο στην νομισματική πολιτική. Όταν ήμουν υπουργό Οικονομικών, διαπίστωσα τις δυσκολίες στο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών. Εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στα εθνικά μας ζητήματα και ξεχνάμε τα άλλα. Όμως η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να ε, αποφεύγουμε τους τριγμούς εξαιτία εξωτερικών ε, σοκ. Και όλα αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία εγώ τα λέω έτσι από το κεφάλι μου. Έχω δουλέψει πάρα πολύ όσον αφορά την απλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των κανόνων που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση και την εμβάθυνση των αγορών. Βραχυπρόθεσμα, μετά τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και με την προστασία που έχουμε από το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και δημιουργώντας επίσης και άλλα δημοσιονομικά εργαλεία θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά. Σε συνδυασμό μάλιστα με άλλες μεταρρυθμίσεις στα συστήματα πληρωμών, αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να υποφεληθεί ακόμα περισσότερο το ευρώ εφόσον αποτελέσει αποθεματικό σε διεθνές επίπεδο και θα μπορέσει να διατηρήσει περισσότερο την ανεξαρτησία του μέσα σε έναν όλο και περισσότερο βέβαιο κόσμο. Η δεύτερη διάσταση της ε, συμμετοχής, όπως έλεγα, είναι η ποικιλομορφία. Ο Πολ Βαλερή είχε πει ότι πρέπει να βάλουμε από κοινού ό,τι καλύτερο έχουμε και να πλουτίσουμε από τις διαφορές μας. Η Σιμών Βέιλ επίσης έκανε μια αντίστοιχη ε, παρατήρηση όταν ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ πιστεύω ότι η ποικιλομορφία αποτελεί πλούτο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε ταλέντο, κάθε γνώση και πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως οφείλου, ε, φιλής, ε, υποβάθρου, προέλευσης και να ακούμε επίσης παντός είδους φωνές όσο γίνεται περισσότερο και να διασφαλίσουμε ότι ο διάλογος αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εκπόνησης πολιτικής. Και γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ για το διάλογο που θα μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας εφόσον επιβεβαιωθώ ω επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να ακούει και πρέπει να καταλαβαίνει τι αγορέ. Δεν πρέπει να την καθοδηγούν οι αγορέ, όχι, αλλά να ακούει και να καταλαβαίνει. Επίση πρέπει να ακούει και να καταλαβαίνει τον κόσμο. Γιατί ένα νόμισμα αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο ανήκει στον κόσμο. Όταν ήμουν στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, δούλεψα σκληρά προκειμένου οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σκληρά και να διασφαλίσουμε ότι οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών και οι άνθρωποι ε, νιώθουν δικό του το νόμισμα αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πιστεύω ότι μόνο αν έχουμε ένα ζωντανό διάλογο μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Συνεπώς, ε, πρέπει να έχουμε τη δέσμευση στις ε, εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χρειάζεται προσαρμοστικότητα και χρειάζεται και συμμετοχή όλων. Χρειάζεται επικοινωνία. Προσβλέπω λοιπόν σε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων μαζί σας και με εδώ μόνο για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Έχω ετοιμαστεί σκληρά έχω την εμπειρία που έχω συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είμαι εδώ για να ακούσω και τις δικές σας τις απόψεις και για να καταλάβω τι εσείς περιμένετε από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, αλλά πρέπει να προσαρμόσουμε και το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Στον πρώτο γύρο ερωτήσεων, πέντε λεπτά για τον καθένα και μετά στον επόμενο γύρο ερωτήσεων θα δούμε πόσο χρόνο θα έχει ο καθένας. Ο κύριος Φέρμπερ, εκ μέρους του ΕΛΚ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα μου επιτρέψετε, ε, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα εξ ονόματος του ΕΛΚ να σα καλωσορίσω θερμά, ε, ενδεχομένω σε μια νέα θέση ε, στην προηγούμενη θέση σα, ε, είχατε έρθει επανειλημμένα, σα είχαμε δει εδώ, με γενικά λόγια μα παρουσιάσετε ποια είναι τα καθήκοντα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και εγώ εκεί θέλω να εστιάσω στην εντολή που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη τελική ανάλυση υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που αποφασίζουν για άλλα θέματα, θέματα όμω που δεν έχουν καμία σχέση με τι αρμοδιότητε τη ΕΚΤ. Εσεί, λοιπόν είπατε ότι πρέπει κανεί να δει το πλωστάσιο των εργαλείων ε, που υπάρχουν την Εγώ διάβασα μία μελέτη που προέκυψε κατά τη διάρκεια τη θυσία σα και εκεί αναφέρεται ότι πρέπει να καταργηθούν οι συναλλαγέ ε, μετρητά. Ε, θα πρέπει επίση ε, να γίνεται σωστό υπολογισμό των υπολείπων εγώ λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα, ε, τι ακριβώς έχετε κατά νου όταν λέτε ότι θα πρέπει κανείς να εξετάσει και νέα καινοτόμα εργαλεία έτσι ώστε να υλοποιήσει την εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Uh, το 2008 και πιο συγκεκριμένα το 2014 πολύ λίγοι άνθρωποι θα περίμεναν να υπάρξουν ε, κάποια εργαλεία ε, ορισμένα εξ αυτών ε, τα ανακάλυψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είτε πρόκειτο για μακροπροληπτικά εργαλεία, είτε πρόκειτο για προγράμματα αγοράς διαφόρων άλλων εργαλείων, είτε πρόκειτο για στοχευμένους ε, μηχανισμούς ε, χρηματοδότησης. Νομίζω ότι ε, τότε κανείς δεν περίμενε ότι πολλοί θα ήταν αναγκασμένοι να καταφύγουν σε άλλα εργαλεία. Έγινε λοιπόν πολλή δουλειά για να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα της εποχής. Και προφανώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εστίασε στο να ανταποκριθεί στο 1.127 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυρίως εστιάζει στην σταθερότητα των τιμών. Έχοντας λοιπόν κατά νου την σταθερότητα των τιμών χρησιμοποιήθηκε ένα οπλοστάσιο ε, έτσι ώστε να έχουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ξέρετε είναι πάντα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τις αντιδράσεις, γιατί σε όταν υπάρχουν συγκεκριμένε αντιδράσει, πρέπει κανεί πάντα να υπολογίζει τι θα γινόταν αν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο. Πάντω, εμεί προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε την αξία όλων αυτών των εργαλείων και είναι σαφέ ε, ότι αυτά τα εργαλεία βοηθούν έτσι ώστε να αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη το 2% είναι εκεί που έφτασε η ΕΚΤ και πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτής της ανανεωμένης εμπιστοσύνης, έχοντας το βλέμμα προς το μέλλον. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι απειλές, ποιες είναι οι συνθήκες, ε, ποια είναι τα πιο κατάλληλα εργαλεία από αυτά που έχουμε και μέσα στο περιθώριο που υπάρχει για να χρησιμοποιηθούν, ε, ποια είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους στην χρήση αυτών των εργαλείων και μέχρι ποιου βαθμού. Πρόκειται λοιπόν σαφώς για αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται ε, συλλογικά από το ε, Προεδρείο μας, από το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Δεν θέλω να πω τι θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου. Ε, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ ενδεχομένω να συμμετέχω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καθορίσω τίποτα. Εγώ Πιστεύω ότι η ανάλυση κόστους ωφέλους και ίσως και η αναθεώρηση ε, του νομισματικού πλαισίου που θα πρέπει να γίνει όχι μόνο από την ΕΚΤ αλλά και σε συνεργασία με, άλλους, με άλλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, αυτό είναι επιτιμητό λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν. Γιώνας Φερνάντες παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Η δική μου η ερώτηση που είχα προετοιμάσει μοιάζει πάρα πολύ με αυτή που έκανε ο κύριος Φέρμπερ, αλλά ίσως με κάποια διαφορετική απόκριση. Ε, στις γραπτές σας απαντήσεις σε αυτήν την Επιτροπή υπάρχει μία απάντηση που δίνεται και θέλω να διευκρινίσετε στην ερώτηση παριθμών 6 σχετικά με την δυνατότητα να προαχθούν ή όχι ε, τα νομισματικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς αναφέρεστε στις ε, αλλαγές ε, που έγιναν από την αρχή της κρίσης, αλλά δεν μας δίνεται μια ξεκάθαρη θετική ή αρνητική απάντηση. Το πλαίσιο υπάρχει από το 2003 πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση και χρησιμοποιήθηκε από την ΕΚΤ ως ένα συμπληρωματικό μέτρο. Έκτοτε όμως ε, ε, μειώθηκαν τα επιτόκια και αυτό ε, προέκυψε στο να μειωθούν και περιορισμοί από τις τράπεζες. Συμφωνώ με τον κύριο Φέρμπερ ότι πρέπει να αυξήσουμε το πραγματικό, όχι το ονομαστικό επιτόκιο. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση νομίζω ότι αξίζει να ε, δούμε λιγάκι το πλαίσιο, να το αναλύσουμε να μελετήσουμε τα περιθώρια που υπάρχουν για την ε, αύξηση του ε, κανονικού, του κανονικού επιτοκίου και θα ήθελα να μας πει τι μπορεί να κάνει η ΕΚ σε περίπτωση πραγματικής κρίσης. Υπάρχουν οι στόχοι που έχουν αναφερθεί ή ενδεχομένως και μελέτη κάποιας, ε, κάποιου ψηφιακού νομίσματος. Εσείς ε, στηρίζετε αυτό το νομισματικό πλαίσιο που έχει στηρίξει παραδείγματο χάρη η Τράπεζα του Καναδά ή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και μπορείτε να είστε λίγο πιο σαφείς από ό,τι στη γραπτή σας απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, στην γραπτή μου απάντηση προσπάθησα να είμαι ε, ουσιαστική να απαντήσω, αλλά θα επανέλθω στη δική σας την ερώτηση. Κοιτάξτε, από το 2003 έχει περάσει πάρα πολύ καιρό και από τότε έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά την ΕΚΤ. Αν δούμε λιγάκι άλλες κεντρικές τράπεζες που είναι αξιοσέβαστες με πολύ καλή φήμη, η Bank of Canada, η Τράπεζα του Καναδά, αλλάζει το ρυθμιστικό της πλαίσιο κάθε πέντε χρόνια. Η Fed των ΗΠΑ ξεκίνησε μία αναθεώρηση του ε, ρυθμιστικού πλαισίου πριν από έξι μήνες και θα διαρκέσει 12 μήνες για να μπορέσει να λάβει υπόψη της όλους τους ενδιαφερόμενους να κάνει απολογισμό όλων των απόψεων που έχουν σχέση με το πλαίσιο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι με την ειν προεδρία του κυρίου Ντράγκη υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία επανεξέτασης κάποιων στοιχείων του νομισματικού πλαισίου. Έχω κατά νου κυρίως αυτά τα οποία ελέγχθησαν τον Ιούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε κατά πόσον ο πληθωρισμός που είναι κοντά ή κάτω από 2% κατά πόσον ο πληθωρισμός θα πρέπει να επιτυγχάνεται από κάτω ή με ένα ασύμετρο τρόπο κατά πόσον αυτός είναι ήδη ένας τρόπος για να ανεθωρηθούν στοιχεία του ε, νομισματικού πλαισίου. Πιστεύω λοιπόν ότι η διευκρίνηση του στόχου είναι κάτι ε, το οποίο έχει ήδη εξεταστεί. Ε, δεν είναι σαφές ακριβώς ποιος είναι ο στόχος. Σε τελική ανάλυση, ε, τι είναι κοντά στο 2%, μιλάμε 1,6 για 1,9. Υπάρχει ευελιξία και εγώ εξ όσων μπορώ να καταλάβω αυτά που μας λέει ο πρόεδρος τουλάχιστον της ΕΚΤ είναι ότι δεν είναι το 1,6. Δεν λέει ακριβώς τι είναι. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν βρεθεί σε αρμοδιότητα κεντρικού τραπεζίτη καταλαβαίνουν πολύ καλά το πόσο λεπτό είναι όλο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήταν ο κεντρικός ε, τραπεζίτης ε, στην Αυστραλία, στο Jackson Hole, εκεί συναντήκαμε όλοι μας και εκείνος είπε ε, Καταλαβαίνει, πιστεύετε κανείς ένας μέσος άνθρωπος γιατί δαπανάμε τόσο πολύ χρόνο που να λέμε κοντά στο 2% αλλά όχι πάνω από τους 2%. Άρα δηλαδή πρώτον πρέπει να διευκρινίσουμε, να ερευνήσουμε, να συνυπολογίσουμε απόψεις, να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις και με βάση ανάλυση κόστους ωφέλους να διευκρινίσουμε καλύτερα το πλαίσιο. Εγώ ε, λοιπόν ενθαρρύνω και στηρίζω αυτήν την εξέλιξη εξέλιξη ε, και βεβαίως χρειάζεται η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για να ληφθεί η περαιτέρω απόφαση. Εκ μέρους του Renew Europe, ο κύριος Λουί Γκαρικάνο. Κύριε Λαγκάρντ, σας εύχομαι καλή επιτυχία με όλη την εμπειρία που έχετε και τι ικανότητε που έχετε για τη νέα θέση στην οποία έχετε οριστεί. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Ο λαϊκισμός και ο εμπορικός πόλεμος ε, που έχει ξεκινήσει από τον πρόεδρο Τραμπ και άλλα σοκ στην παγκόσμια οικονομία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε νέα ύφεση. Αυτό που με απασχολεί και εμένα προσωπικά και πολλούς Ευρωπαίους πολίτες είναι ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι προκατοχοί σας εξήγησαν ή σχεδόν εξήγησαν τα συμβατικά μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερο πεδίο για χαμηλότερα ή πολύ χαμηλότερα επιτόκια ή για ε, συνέχιση αυτής της νομισματικής πολιτικής. Πολλοί διερωτώνται αν υπάρχει περαιτέρω περιθώριο. Όσον αφορά την Ευρωζώνη, δεν έχουμε κάνει όλα όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχουν γίνει πολλά διαρθρωτικά ε, ζητήματα πολλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει, δεν έχουμε ένα δημοσιονομικό εργαλείο για σταθεροποίηση της οικονομίας, πολλά δεν έχουν γίνει. Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι δύο στους δύο αυτούς τομείς. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να καταπολεμήσει μια πιθανή νέα ύφεση. Σε αυτή την περίπτωση, τι εργαλεία χρησιμοποίησε στο παρελθόν, τι νέα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Και δεύτερον, για την Ευρωζώνη έχει κάνει η Ευρωζώνη ότι μπορούσε να κάνει μέχρι τώρα. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. ποιε είναι οι δικέ σα προτεραιότητε, Τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να κάνει το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και πώ βλέπετε το δικό σα ρόλο στο να προωθήσετε αυτά τα οποία πρέπει να κάνει η Ευρωζώνη. Είτε πρόκειται για ασφάλιση καταθέσεων, είτε μηχανισμό ασφαλείας, διάσωση. Ευχαριστώ. Κύριε Λαγκάντε, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια στην αρχή. Θυμάμαι στην εποχή της κρίσης, πολλοί διοικητές κεντρικών τραπεζών ε, διαμαρτύρονταν ε, λέγοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να δώσει λύση. Και βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι διοικητέ κεντρικών τραπεζών χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν στην εργαλειοθήκη τους, ε, χρησιμοποιούν και επανεξετάζουν όλες τι πολιτικές κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα διαθέσιμα εργαλεία και αυτό πρέπει να κάνουν σύμφωνα με την ε, εντολή που έχουν. Σαφώς ε, πρέπει να υπάρχει συνεργασία και όλα τα θεσμικά όργανα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη συγκεκριμένα για να ανταποκριθούμε στις απειλές ε, του λαϊκισμού πρέπει να υπάρξει τέτοια συνεργασία. Ε, όταν και αν γίνω πρόεδρος ε, της ε, ΕΚΤ υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε για το ρόλο που μπορούν να παίξουν πολλές χώρες. Το έχω πει πολλές φορές ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι ορισμένες χώρες στην Ευρωζώνη μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημοσιονομικό χώρο που έχουν για να βελτιώσουν τις υποδομές, τις τα ευρωζωνικά δίκτυα, να καταπολεμήσουν δηλαδή ε, τις πηγές ύφεση. Και υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες σήμερα. Αν δείτε τις χώρες της ευρωζώνης, αν δείτε τις χώρες που βρίσκονται περίπου σε μηδενικό έλλειμμα ή με 0,5% έλλειμμα, οι περισσότερες χώρες στην Ευρωζώνη είναι σε αυτή τη θέση. Άρα, σαφώς δεν υπάρχει μεγάλο πεδίο, αλλά υπάρχει πεδίο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις δημοσιονομικές πολιτικές. Δεύτερον, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε πάρα πολλές χώρες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σε μερικές χώρες έχουν ξεκινήσει, κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, έχουν εξεταστεί χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα όμως και σαφώς οι χώρες που δεν έχουν το δημοσιονομικό χώρο σήμερα, λιγότερο από το ίμιση των χωρών της Ευρωζώνης, πρέπει να επανασχεδιάσουν ε, το μείγμα δημοσιονομικών πολιτικών και πολιτικών υπέρ της ανάπτυξης, ε, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτές είναι οι συνθήκες στις οποίες μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις καλύτερα και να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα τώρα που υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Το σωστό μείγμα λοιπόν κατάλληλης νομισματικής πολιτικής με όλα τα διαθέσιμα μέσα, νομισματικές, ε, δημοσιονομικές συγγνώμη, πολιτικές με τις χώρες που μπορούν ε, να τις χρησιμοποιήσουν και διορθωτικές μεταρρυθμίσεις παράλληλα. Σβέν Γκίγκολ, εκ μέρους των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ. Κυρία Λαγκάρντ, καταρχήν θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, για την οποία είστε υποψήφια ε, να γίνεται πρόεδρο. Είναι μια, ένα, ένα θεσμικό όργανο ιδιαίτερα ισχυρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι καλό μήνυμα, καλό ιονό το ότι μια ισχυρή γυναίκα θέτει υποψηφιότητα για ένα ισχυρό οργανισμό και θα ήταν καλό αυτό ο ισχυρό οργανισμό ε, να έχει επικεφαλή μια γυναίκα. Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από άνδρες είναι καλό να έχουμε γυναίκε υποψηφίου για τέτοιε θέσει. Πέραν τούτου θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που έσωσε το ευρώ και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Όχι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, αλλά η ΕΚΤ έσωσε το ευρώ. και μετά την νομισματική πολιτική ε, επήλθε ένα ε, επίπεδο λαϊκισμού πάρα πολύ υψηλό οι πολιτικοί δεν έκαναν τη δουλειά τους και χρειάστηκε από την ΕΚΤ παρέμβαση για στενότερη συνεργασία, για δημιουργία ενιαίας αγοράς και καλύτερη συνεργασία στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που η ΕΚΤ έπρεπε να είναι επιθετική στη νομισματική της πολιτική. Και το είπατε κι εσείς ότι τα βλέπετε τα προβλήματα, βλέπετε τις ανησυχίες των πολιτών λόγω των αρνητικών παρενεργειών της επιθετικής πολιτικής είχα την εντύπωση ότι ο προκάτοχός σας δεν επικοινωνούσε με όλους τους πολίτες, δεν προσπαθούσε να εξηγήσει με πιστικό τρόπο γιατί απαιτούνται αυτά τα μέτρα που λαμβάνονταν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες είδατε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους πολίτες και να εξηγήσετε τις αρνητικές επιπτώσεις. Αναφέρεται επίσης και το πρασίνισμα της χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρχει χρηματοπιστωτική και νομισματική σταθερότητα χωρίς καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και η ΕΚΤ πρέπει να παίξει το ρόλο της γιατί είναι το πιο ισχυρό χρηματοπιστωτικό όργανο. Στι απαντήσει σα λέτε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να το κάνει. Δεν είναι αρκετά ισχυρή η διατύπωση στην απάντησή σα. Μπορείτε να είστε πιο στεναροί και πιο τολμηροί σε αυτό το πρασίνισμα της χρηματοπιστωτικής πολιτικής υπό την ηγεσία σας στην ΕΚΤ απάντηση. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω την προσωπική μου θέση για το θέμα αυτό και το κάνω με προσοχή γιατί δεν θέλω με αυτά που λέω να δεσμεύσω το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γιατί εγώ απλώς ε, είμαι υποψήφια για τη θέση, δεν είμαι πρόεδρος της ΕΚΤ. Η προσωπική μου θέση για αυτά τα θέματα είναι ότι σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο οι κίνδυνοι για από την κλιματική αλλαγή ε, και για την προστασία του κλίματος πρέπει να βρίσκονται ως βασική προτεραιότητα. Βεβαίως σταθερότητα, αλλά θα πρέπει ε, και η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι για το περιβάλλον να θεωρούνται βασική αποστολή όλων των θεσμικών οργάνων. Και πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το, το σπίτι του ο καθένας για να μπορέσει να προχωρήσει και πιο πέρα να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό ίσχυε και όσο ήμουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα μιλήσω για το ΔΝΤ πριν μιλήσω και για την ΕΚΤ. Κλιματικός κίνδυνος λοιπόν, αλληλεγγύε για το περιβάλλον και το δημοσιονομικό τμήμα και πολλά άλλα τμήματα, πολλές άλλες διευθύνσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επικέντρωσαν την προσοχή τους σε ε, ενισχύσεις που δίδονταν, παραδείγματος χάρη για τα ορυκτά καύσιμα, το άμεσο και το έμεσο κόστος αυτών των ενισχύσεων. Επικεντρωθήκαμε επίσης ε, σε προπολογισμού που θα έπρεπε να είναι δημοσιονομικά υπεύθυνοι. Αυτά για το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Τώρα για την ΕΚΤ, χωρί να προδικάζω τι μπορεί να συμβεί, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τελικά υπό την ηγεσία ε, του ε, Προέδρου. Και πάλι, όπω και στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, έτσι και για την ΕΚΤ, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ίδιο μα ε, τον οργανισμό για να ληφθούν οι αποφάσεις ε, για το πού θα επενδύσει ο κάθε οργανισμός και για το πρασίνισμα του δικτύου. Όταν υπάρχουν οι διοικητέ κεντρικών τραπεζών ε, που λένε ότι οι αλλαγέ ε, στο κλίμα είναι βασική κίνδυνη που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες. Αν το άκουγα αυτό ω τράπεζα θα ανησυχούσα και θα άρχιζα να κοιτάζω τι προβλέψει μου. Θα άρχιζα να επανεξετάζω το, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Όσον αφορά τις επενδύσεις, και δεν θα μακρηγορήσω, η ΕΚΤ δεν μπορεί αποκλειστικά και μόνο να επενδύει. 2,6 δισεκατομμύρια χαρτοφυλάκιο δεν μπορεί να επενδύει αποκλειστικά σε πράσινα ομόλογα διότι δεν ε, υπάρχουν αρκετά ε, στην αγορά. Αλλά αν δώσει ε, μηνύματα ότι θα μπορέσει να επενδύσει και η αγορά θα το καταγράψει και επομένως οι κατευθύνσεις των επενδύσεων θα έχουν κάποια ένδειξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Έχω μία ερώτηση. Αναφερθήκατε λίγο στην αρχική σας παρουσίαση. Πολλά υπόθηκαν για τον πολυμερή κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε και έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο επιθετικές αυτοκρατορίες την Αμερικανική με το δολάριο και την ε, Κινέζικη που προσπαθούν να επιτεθούν και μία και άλλη. Λοιπόν, στις διεθνείς συναλλαγές, τι εργαλεία έχουμε οι κεντρικές τράπεζες. Δεν θα έπρεπε να είχαμε κάτι υπέρ της ανεξαρτησίας των χωρών μελών. Και στα πλαίσια της εντολής σας, πώς φαντάζεστε, τι φαντάζεστε ότι θα κάνετε προκειμένου το ευρώ να γίνει διεθνές νόμισμα, ε, για τις συναλλαγές ή ως ε, αποθεματικό όπως θα έπρεπε να είναι και πώς το τραπεζικό σύστημα ε, θα είναι αντοχής για να μπορεί να αποφύγει τις επιθέσεις αυτές των αυτοκρατοριών. Είχα και μια άλλη ερώτηση, την οποία βέβαια σε ένα μεγάλο μέρος απαντήσατε. Εγώ θεωρώ ότι η αξιοπιστή ενός νομισματικού συστήματος εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό το σύστημα και στις ικανότητές του να ανταποκριθεί στις ε, προσδοκίες. Είναι ξεκάθαρο όμως και το είπατε και εσείς, η περιβαλλοντική κρίση τελικά και οι αντιπαραθέσεις στην ανθρωπότητα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Η αξιοπιστία πάντως του νομισματικού συστήματος με τι εργαλεία θα εξασφαλιστεί για να ξεπεράσουμε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Η κυρία Λακάρδη, ευχαριστώ για την διτή αυτή ερώτηση. Για την πρώτη σας ερώτηση για το ευρώ. Ένα νόμισμα για νομισματικά αποθέματα και διεθνές νόμισμα να αναγνωριστεί έτσι και πώς θα κρατήσει τη θέση του ανάμεσα σε δύο αυτοκρατορίες που αντιπαρατίθεται αυτή την εποχή. Μα το ευρώ ήδη σήμερα είναι ένα νόμισμα στο οποίο υπάρχουν μεγάλα αποθέματα. Παρά τις όποιες προσπάθειες κάνουν άλλες κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές, το δολάριο είναι το πρώτο, αλλά και αυτό αλλάζει. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πρέπει να προσφέρουμε στο ευρώ ε, τα μέσα που χρειάζεται ώστε να είναι πραγματικά ένα διεθνές νόμισμα και για πληρωμές αλλά και για καταθέσεις. Τα συστήματα πληρωμών πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματικά. Επίσης, οι ευρωπαϊκές κεφαλαγορές επίσης θα πρέπει να είναι περισσότερο αναπτυγμένε από ό,τι είναι σήμερα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρόεδρο Γκουαλτιέρη, γιατί ξέρω ότι έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην ενίσχυση και στην ευάθυνση των κεφαλαγορών στην Ευρώπη αγορά κεφαλαίων που δεν είναι θέμα βέβαια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί βασικό στοιχείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αν πολλαπλασιάσουμε τις πηγές χρηματοδότησης για όλους τους οικονομικούς φορείς και αν προσφέρουμε εναλλακτικέ στα τραπεζικά συστήματα, ενισχύουμε το ρόλο του ευρώ. Και υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε αλλά είναι πιο μακροπρόθεσμο, είναι να έχουμε στη διάθεσή μας ένα μέσο, γιατί έχουμε το Αμερικανικό θησαυροφυλάκιο που εξασφαλίζει αυτούς που ανησυχούν. Κάτι αντίστοιχο δεν έχουμε σήμερα στην Ευρώπη με αρκετό μέγεθος και αρκετό βάθος για την Ευρωζώνη που να είναι ε, να αντιστοιχεί στο μέγεθος της Ευρωζώνης. Τα μέσα πληρωμή είναι εξαιρετικά αυτά που διαθέτουμε, αλλά πρέπει να τα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο για τις κεφαλαιαγορές και για την ενίσχυση του οπλοστασίου που διαθέτουμε. Απλοποίηση, αποτελεσματικότητα ε, δημοσιονομικών πολιτικών που να είναι συντονισμένες μεταξύ τους, τραπεζική ένωση, ε, μηχανισμός ε, προστασίας καταθέσεων. Όλα αυτά θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το ρόλο του ευρώ ως ε, νόμισμα στο οποίο μαζεύονται καταθέσεις. Κάποιος ο οικονομολόγος έλεγε ότι όλα αυτά γίνονται πολύ αργά μέχρι κάποια στιγμή που ξαφνικά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε τέτοιου είδου εξελίξεις. Ευχαριστούμε. Τώρα για το ECR, ο κύριος Σέπινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω την ερώτησή μου στα Ολλανδικά, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να μάθω για τα αρνητικά επιτόκια. Είναι σαφές ε, ότι η κυρία Λαγκάρτ ακόμα δεν έχει οριστεί βέβαια επικεφαλής, οπότε αφήνει όλες τις εναλλακτικέ ανοιχτές. Όμως τι σημαίνει για τους αποταμιευτές, τους καταθέτες, τους συνταξιοδοτούμενους τα αρνητικά επιτόκια. Γιατί με αρνητικά επιτόκια καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν υπάρχει κάποιος πληθωρισμός. Και έπειτα πρέπει να δούμε και την κλιματική πολιτική. Οι αποταμιευτές είναι στριμωγμένοι στη γωνία, είναι θυμωμένοι, χάνουν. 3% σε 10 χρόνια έχουν χάσει το 1 τρίτο του κεφαλαίου τους, που εξαφανίζεται, εξατμίζεται. και αν αυτά όταν έχουμε μηδενικό επιτόκιο, όταν αρχίσουμε με τα αρνητικά επιτόκια τι θα γίνει. Ο κόσμος θα γυρίσει ανάποδα. Ξαφνικά θα γίνεται η βασίλισσα του ευρώ. Όμως φοβάμαι ότι με τα αρνητικά επιτόκια θα έχετε εναντίον σας ε, τους ε, ανθρώπους στο δρόμο. Οι αποταμιεύσεις πρέπει να επιβραβεύονται και όχι το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Δεν μιλάω Ολλανδικά, δυστυχώς, οπότε θα σας απαντήσω αγγλικά. Νομίζω ότι στην ερώτησή σας έχω δώσει δύο απαντήσεις νωρίτερα, απαντώντας άλλους. Πάντα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση κόστους-οφέλους για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τον ε, πολλαπλή ρόλο του πληθυσμού Κάποιοι είναι δανειστές, κάποιοι δανείζουν, κάποιες χώρες μέλη είναι βαριά χρεωμένες, κάποιες άλλες όχι. Και οι επιπτώσεις του όποιου επιτοκίου εξαρτάται από το για ποιον μιλάμε. Όταν λοιπόν αναθεωρούμε το πλαίσιο και εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των μέσων που έχουμε χρησιμοποιήσει, πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλους αυτούς τους ρόλους τις διαφορετικές περιπτώσεις και να αποφασίσουμε σε τι βαθμό και πόσο βαθιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια μέσα για να έχουν καθαρά θετικό αποτέλεσμα. Αν υπάρχει ύφεση, αν υπάρχει το αντίθετο, εξαρτάται από τον ε, στόχο κάθε φορά και μην ξεχνάμε ότι αν διαπιστώσουμε ότι δεν είναι καλό για τον κόσμο, θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή. Πάντως, η νομισματική πολιτική με την προσφορά χρήματος είναι κάτι που χρειάζεται και θα χρειάζεται ακόμα για κάποιο καιρό. Και αυτό βέβαια χωρίς να ξέρουμε τι θα αποφασίσει τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα προς το παρόν. Και επιτρέψτε μου, γιατί έχω ένα λεπτό που θέλω να το χρησιμοποιήσω ακόμα. Πολύ σύντομα. Γι' αυτό που λέτε για τα θετικά και τα αρνητικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσω να βοηθήσω να κοινωνήσω το λόγο, το στόχο που προσπαθώ να πετύχω. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Όχι αγορές, γιατί αγορές καταλαβαίνουν όλες τις γλώσσες, όλα τα αρχικά που συζητάμε και πετάμε δεξιά και αριστερά. Όχι. Ο κόσμος της Ευρωζώνης πρέπει να καταλάβει γιατί παίρνονται αποφάσεις που παίρνονται. Ποιο είναι το θετικό, ποιος είναι ο απότερος στόχος, ε, ποια θα είναι η ζημιά στην αρχή και το ωφέλει αργότερα. Σε αυτά τα πράγματα θέλω εγώ να σπαταλήσω ενέργεια και χρόνο. Τελευταία σε αυτόν τον πρώτο κύκλο. Κυρία Μανώ ε, Καλημέρα. Επανέρχομαι μετά την παρατηρήση του Σβέν. Όταν ε, ε, ομιλώ πρώτη γυναίκα ομιλήτρια, μπορώ κι εγώ να πω ότι είναι κρίμα που δεσπόζει η αντρική παρουσία σε τέτοιους τομείς. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για δύο βασικά θέματα την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η νομισματική πολιτική παίζει θεμελιώδη ρόλο για αυτά τα δύο θέματα. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Ε, δούλευα μέχρι τώρα για μία μη κυβερνητική οργάνωση, την Oxfam, που είχε ως βασικό αντικείμενο την καταπολέμηση των ανισοτήτων και χρησιμοποιούσαμε ε, τις ε, δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα θέματα ανισοτήτων. Και πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας το ερωτηματολόγιο απογοητεύτηκα κάπως γιατί βλέπω ότι η λέξη ανισότητα μόνο δύο φορές εμφανίζεται, ενώ η σταθερότητα των τιμών εμφανίζεται 28 φορές. Ε, ίσως στις απαντήσεις σας μας δίνετε και την εικόνα των προτεραιοτήτων σας. Πάνω από χίλια δις έχουν δοθεί στο ε, τραπεζικό σύστημα και ε, μόνο 230 ε, σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά. Τεράστια ποσά δόθηκαν σε τράπεζες, βοηθώντας την κερδοσκοπία στις χρηματαγορές. Και ο Μάριο Ντράγκη είπε ότι οι πλέον πλούσιοι επωφελούνται κατά πάσα από, το, από την ποσοτική χαλάρωση. Ε, τι συγκεκριμένα μέτρα είστε πρόθυμοι να πάρετε για να βελτιώσετε την πραγματική οικονομία ώστε να μην επιδεινωθούν οι ανισότητες. Ο στόχος του να περιοριστεί ο πληθωρισμός που δεν είναι πλέον προσαρμοσμένος στην οικονομική συγκυρία με χαμηλή ανάπτυξη και πληθωρισμό ε, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ε, φούσκα της κερδοσκοπίας που είδαμε τα τελευταία χρόνια και πώς μπορούμε να ενσωματίσουμε και άλλες παραμέτρους και όχι μόνο τη σταθερότητα των, των τιμών. Ε, χαίρομαι για αυτά που διάβασα στο ερωτηματολόγιο, στις απαντήσεις που δώσατε. Μιλάτε για την πράσινη συμφωνία. Ε, και εδώ θέλω να κάνω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι πώς μπορούμε να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε τις μορφές ενέργειας που ρηπαίνουν γιατί ο ιδιωτικός δανεισμός ε, έχει ωφελήσει κυρίως επιχειρήσεις που ρηπαίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό και δεν λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια στη χρηματοδότηση της ΕΚΤ θα μας μιλήσετε για τα πράσινα ομόλογα, αλλά και εσείς θα αναγνωρίζετε ότι είναι περιορισμένο το μέγεθος της αγοράς και δεν πρέπει και να στρεβλώσουμε την αγορά. Επομένως, εδώ έχουμε και ένα παράδοξο. Και άλλο ένα ερώτημα, πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η οικολογική παρέμβαση, αυτή η μετάβαση προς μια πιο, ένα πιο οικολογικό μέλλον. 190 δις το χρόνο χρειάζονται για τη χρηματοδότηση. Μιλάτε και για το ρόλο του δημοσίου τομέα και τη δημόσια χρηματοδότηση. Στη σελίδα 26 λέτε κάτι που μου με εξέπληξε, ότι τελικά η νομισματική πολιτική δεν είναι πανάκια, δεν είναι η βασική πολιτική για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Πώ μπορεί να αναπροσαρμοστεί η νομισματική πολιτική για την προοπτική τη κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Για την ερώτησή σας σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων, όντως είναι ένας τομέας ε, στον οποίο αναλάβαμε δεσμεύσεις ε, στο Δουνουτού και δουλέψαμε πολύ με την Oxfam ε, με φίλους με τους οποίους προσπαθήσαμε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και για, τα δύο, και για τους δύο οργανισμούς, και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για την Oxfam. Είναι σαφές ότι η σταθερότητα των τιμών παραμένει η βασική έδρα της ΕΚΤ, το άρθρο 27 το λέει, το αναφέρει ως πρωταρχικό στόχο. Υπάρχει και δευτερεύον στόχος ε, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι απαραίτητα δευτερεύον γιατί μόλις έχουμε σταθερότητα των τιμών, μόλις το επιτύχουμε θα δούμε ποιοι είναι και ε, οι στόχοι των άλλων θεσμικών οργάνων ώστε να έχουμε κάποια εναρμόνιση. Ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί επομένως απολύτως να αποτελέσει στόχο και της ΕΚΤ στις πολιτικές της. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για την απάντησή μου σχετικά με το πρασίνισμα και το πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη. Τα πράσινα ομόλογα όντως ε, είναι μικρά σε αριθμό και νομίζω ότι η ΕΚΤ ε, μέχρι τώρα έχει παίξει κάποιο ρόλο. Υπάρχει και ένα πολύ καλό ε, έγγραφο επί του οποίου θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Πρέπει ε, να καθοριστεί τι αποτελεί πράσινη επένδυση και τι όχι. Μέχρι τώρα υπάρχει ταξινόμηση σε πολλά επίπεδα, αλλά χρειάζεται μια διευκρίνηση του τι ακριβώς ε, εννοούμε και η ΕΚΤ που κάνει δράσεις αναχρηματοδότησης ε, προϊόντων που φτάνουν σε περίοδο ρήμανσης θα δώσει τη δυνατότητα ε, να αλλάξει κατεύθυνση και να κατευθυνθεί προς ε, πιο πράσινα προϊόντα. Θα συνεχίσω λοιπόν να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα για να μπορούμε πώς η ΕΚΤ μπορεί να δράσει. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος και για να υπάρχει κάποιος βαθμός ισότητας για όλους τους βουλευτές θα ήθελα να βάλουμε ένα όριο 4,5 λεπτών και παρακαλώ κάνετε σύντομες ερωτήσεις. Ο κύριος Ότμαρ Κάρας. Κυρία Λαγκάρτ, σας συγχαίρω για την, για την πρόταση ορισμού. Για μένα ε, το θέμα της ECB, της ΕΚΤ, ε, δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί, είναι κάτι που αποτελεί μέρος του προβλήματος. Εσείς ε, εξηγήσατε τις προκλήσεις που υπάρχουν. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε την παγκόσμια προοπτική σας. Η επιτυχία σας στη θέση της Πρόεδρου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και η συμμετοχή σας στους G20 και στα προγράμματα οικονομικής στήριξης σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στην Τρόικα, όλα αυτά σας ενίσχυσαν και σας ενισχύουν στη θέση της υποψηφίου του ΕΚΤ. Κάποιοι πολιτικοί όλο και περισσότερο ε, λένε ότι η ΕΚΤ φταίει για πάρα πολλά δεινά, ε, η ΕΚΤ φταίει για την αποτυχία, επικρίνουν το χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων. Αυτή η κριτική ε, προσκρούει σε ότα και θέλω να σας ρωτήσω πώς ακριβώ σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το έλλειμμα. Those are very broad questions. Thank you. Η ερωτήσεις σας καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα. Ε, κοιτάξτε, το να γίνω πρόεδρος της ΕΚΤΑ, αυτό σημαίνει ότι θα φέρω μαζί μου και την εμπειρία που έχω συγκεντρώσει σε διάφορες θέσεις. Και αυτό που βίασα στους ε, G20, στις διάφορες αντίσεις των G7, όλα αυτά που διαπίστωσα είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε αυτές τις ομάδες, οποτεδήποτε εμφανίζονται και ακραίες προκλήσεις. Ε, βεβαίως δεν επιτιμώ να υπάρχουν τέτοιου είδους προκλήσεις, γιατί εγώ αναμφίβολα δεν επιθυμώ ε, να υπάρξει οικονομική κρίση απλά και μόνο για να δείξουμε ότι οι G20, η G7 ε, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εκείνο όμως ε, που θέλω είναι να συμβάλλω σε αυτό το αίσθημα του επίγοντος ε, παρότι αυτή τη στιγμή δεν πληττόμεθα από κρίση. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα του κατεπίγοντος θα συνεχίσει η αναβολή, η αναβλητικότητα και δεν το λέω αν θέλετε με τη μορφή κριτικής αλλά αυτό προκύπτει από τις πολιτικές εκλογές. Ε, οι άνθρωποι καταφεύγουν στο δικό τους το γνώριμο περιβάλλον, στα εθνικά τους συμφέροντα. Ε, περιορίζεται ο δημοσιονομικό του ή ο νομισματικό του ορίζοντα και πιστεύουν ότι κάποιο άλλο θα βρεθεί για να κάνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει. Ε, Έχοντα υπάρξει λοιπόν σε διάφορε θέσει ω υπουργό Οικονομικών, ω επικεφαλής του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που προσπάθησα να εντοπίσω καλύτερη νομοθέτηση, καλύτερα μείγματα πολιτικής, ε, θέλω να πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα καλύτερη συνεργασία, να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτεραιότητες ε, των διαφόρων παικτών και ξέρετε δεν είμαι κάτι το εξοκοσμικό, όπως ίσως κάποιος υπενήχθηκε ε, προηγουμένως, αλλά και εγώ θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα είναι συλλογικά. Είτε μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, για την χρηματοψηφιακή σταθερότητα, την κυβερνοαπειλή, ε, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τη φορολογία, την ε, πολιτική ανταγωνισμό. Όλα αυτά πλέον είναι διεθνή γιατί η πραγματική οικονομία έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο της διεθνικότητας. Και για να ανταποκριθεί κανείς το αίσθημα των πολιτών ότι η μοίρα τους δεν βρίσκεται πια στα χέρια τους και ότι οι εθνικοί ταγοί δεν μπορούν και αυτοί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Και νομίζω ότι το κοινοβούλιο Κοινοβούλιο ε, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Ο κύριος Μαρκές από τους σοσιαλδημοκράτες. Καλημέρα σας κυρία Λαγκάρτ. Η νομισματική πολιτική αποδείχθηκε ότι είναι καθοριστική σημασία για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης, ε, το 2012 ε, είπε ο κύριος Ντράγκη ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των, ε, του δημόσιου χρέους. Αυτό αφορούσε και μια χώρα σαν τη δική μου, την Πορτογαλία. Εσείς θέλω να σας ρωτήσω, αν τελικά εκλεγείτε πρώτος της ΕΚΤΕ και εσείς ε, θα παραμείνετε σε αυτό το δόγμα ότι θα κάνω ό,τι πρέπει πάση θυσία για να διαφυλάξω το ευρώ. Ίσως να χρειαστεί να εφαρμοστούν και αντισυμβατικές πολιτικές για να διαφυλαχθεί το ευρώ και ε, θεωρώ ότι πρέπει ε, για να επιτύχουμε το στόχο μας να ολοκληρώσουμε και το θεσμικό πλαίσιο. Το λέτε αυτό στις απαντήσεις σας. Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, η Τραπεζική Ένωση, ε, κυρίως το ΕΝΤΙΣ, Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα της Ασφάλισης των Καταθέσεων, το ΕΝΤΙΣ. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω όσον αφορά την τα δημοσιονομικά στην Ευρωζώνη. Ε, τι ακριβώς ε, μέτρα προτίθεστε να λάβετε και αυτό που είναι πιο κρίσιμο για τη σταθεροποίηση, θέλω να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να στηρίξετε ένα εργαλείο όπως ε, αυτό που στηρίζει ο η πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, δηλαδή ένα σύστημα για την ε, χορήγηση επιδομάτων, ανεργίας. Εσείς συμφωνείτε σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ και τον προτέρων για την απάντησή σας. Ναι, ο πρόεδρος θα μου πει ότι εσείς το φάγατε το χρόνο και εγώ δεν έχω χρόνο να απαντήσω. Όταν ο πρόεδρος Ντράγκη είπε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σώσουμε το ευρώ και πιστέψτε με αυτά που θα κάνουμε αρκούν, ήμουν παρούσα. Ελπίζω να μην, με, να μου συμβεί εμένα, αλλά αν μου συμβεί θα το κάνω και εγώ. Γιατί πιστεύω ότι οι υπόλοιποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Επιπλέον θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν είπε ότι ό,τι και να χρειαστεί θα το κάνουμε, τελικά αυτό που σχεδιάστηκε ήταν το OMT που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Αυτό που προέκυψε είναι η σταθεροποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ε, να μην είναι δυνατόν να παραλύει ο μηχανισμός ε, μέσα από άλλες εξωτερικές επιδράσεις, γιατί εγώ έχω κάνει την εμπειρία ότι όταν, φτιάξαμε την, ε, όταν προέκυψε η κρίση, να αντιμετωπίσαμε με, τα, με τους διάφορους θεσμούς που φτιάξαμε, ε, τότε δεν ανταποκριθήκαμε αρκετά γρήγορα. Αλλά αν τελικά εκλεγώ, εγώ θα προσπαθήσω να ασχοληθώ κυρίως με την σταθερότητα των τιμών. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά παρακλάδια, πολλές ε, προεκτάσεις ε, για να έχουμε μια σωστή πολιτική. Ως εκ τούτου θεωρώ και να σας πω ε, σχετικά με τις δημοσιονομικές μας αρμοδιότητες. Εμείς από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό που αναγνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα σε κάποια κράτη-μέλη, μεταξύ τους τα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά τι ακριβώς εννοώ. Και η δική μας πρόταση είναι ότι μπορεί κανείς να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να υποβάλει αυστηρά stress test, να δεχτεί ένα εντονότερο βαθμό εποπτείας και έτσι λοιπόν το σύστημα εξασφάλισης καταθέσεων να ισχύει στο σύνολο της ε, Ευρωζώνης χωρίς κανένα περιορισμό. Το ισχύει και για τη δημοσιονομική ικανότητα. Ε, εάν πρέπει να προχωρήσει περισσότερο και εκεί θα πρέπει να υφίστανται οι προϋποθέσεις που θα εγγυώνται ότι αν κάποιος καταθέσει τα χρήματά του σε μία χή χώρα, η χώρα αυτή ε, θα μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα σοκ, βεβαίω στο βαθμό που αυτή, αυτό το σοκ δεν είναι ενδυμικό. Ο κύριος Πασκαλ Καλφά. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ρωτήσω για την σχέση των δικό σας αρμοδιοτήτων και την κλιματική αλλαγή. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς αναφερθήκατε στις αναλύσεις του Μπένου Ακερέλ, που είναι τώρα κεντρικός τραπεζίτης, και είναι ήδη στην εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, το θέμα με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, σταθερότητα τιμών. Αν υπάρξει αλλαγή στο κλίμα 3-5 βαθμοί, σίγουρα θα υπάρξει αλλαγή και στις τιμές. Και επίσης είναι και το θέμα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο Μακερνή και άλλοι τα έχουν πει ότι σήμερα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μεσοπρόθεσμα χρηματοπιστωτική σταθερότητα αν δεν λάβουμε υπόψη μα το θέμα της κλιματικής αλλαγή. Οι δύο ερωτήσεις μου. Πρώτον, δεσμεύεστε να χρησιμοποιήσετε την ταξινόμηση των επενδύσεων και του ενεργητικού σε πράσινα και μη πράσινα και να το λάβετε υπόψη σα. Δεύτερον, αναφερθήκατε στον απολογισμό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, όσον αφορά ε, τα πράσινα ομόλογα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το κάθε ενεργειό και κάθε αγορά που έχει γίνει έχει να κάνει με τον άνθρακα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για πράσινε επενδύσει. Οπότε εσεί μπορείτε να μα πείτε ότι σιγά σιγά η ΕΚΤΕ θα αποδεσμευτεί από αυτό το ενεργητικό το οποίο είναι στεδεμένο άμεσα με τον άνθρακα και τρίτον, θα λάβετε υπόψη σας περισσότερο στις ε, μακροαναλύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το θέμα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα, ελπίζω η ταξινόμηση των επενδύσεων που συζητάτε σήμερα θα καταλήξει σύντομα γιατί πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένα βασικό στοιχείο που σήμερα αποτελεί τροχοπέδι σε διάφορα θέματα, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχω συμμετάσχει σε διάφορα φόρουμ, συζητήσει και με τον ιδιωτικό τομέα και με μεγάλους επενδυτέ, Βρίσκονται σε αβεβαιότητα όσον αφορά την ταξινόμηση αυτή την ιεράρχηση των προϊόντων σε πράσινα και λιγότερο πράσινα. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν ολοκληρωθεί η ταξινόμηση αυτή, τόσο το καλύτερο. Και όπω ε, και εσεί όταν για πρώτη φορά φτάνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι και εγώ είμαι αρχάρια για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, χρησιμοποιεί, θα χρησιμοποιήσει την ταξινόμηση αυτή στο μέλλον. Έτσι εκ προημίου δεν βλέπω γιατί να μην τηρήσει αυτό τον κανόνα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μου φαίνεται προφανές. Τώρα η σημερινοί βέβαια παράγοντες και φορείς θα μου πούν «Α, όχι, ουδετερότητα». Ναι, αλλά αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει μια τέτοια ταξινόμηση, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ουδετερότητα. Θα υπερισχύει η ταξινόμηση δική σας στην ουδετερότητα. Τώρα για το μέγεθος του ενεργητικού, των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον άνθρακα. Ε, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, εννοείται. Αλλά το να πάμε σταδιακά ώστε να απαλείψουμε αυτού του είδους το ενεργητικό που συνδέεται με τον άνθρακα, ε, πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Είμαι πεπισμένη. Αν είμαστε πεπισμένοι για την απόλυτη αναγκαιότητα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο δεσμικό όργανο και αν βρισκόμαστε για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να το κάνουμε. Και προσθέτω και κάτι ακόμα. Στην ανάλυση κινδύνου που κάνουν οι κεντρικές τράπεζες πρέπει στην εποπτική τους αρμοδιότητα να λάβουν υπόψη τους και την κλιματική διάσταση, την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι αποτελεί ένα μοχλό που δεν πρέπει να παραβλέψουμε όταν μιλάμε για προμήθειες, όταν μιλάμε για την εκτίμηση κινδύνου, οι τράπεζες πρέπει να το λάβουν υπόψη τους όταν προσδιορίζουν το κεφάλαιό τους. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, Διαφερέιρα, από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Λαγκάρτ, είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μια γυναίκα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι η πρώτη φορά που η εντολή της ε, Τράπεζας και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκινούν συγχρόνως. Είναι καλό. Όταν θα έχετε εκλεγεί θα μπορέσετε να συνεργαστείτε μεταξύ σα για να προχωρήσει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση που αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε. Τώρα, στην τελευταία τη συνεδρία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούλιο αναφέρθηκαν μέτρα για την τόνωση τη ευρωπαϊκή οικονομία. Και κάποια μέλη τότε μίλησαν ενδεχομένω για ένα πακέτο μέτρο, όπως μείωση επιτοκίων και αγορά ενεργητικού. Τον Μάρτιο στην Πορτογαλία είπατε ότι πρέπει να αυξήσουμε την προσπάθεια για την μείωση του χρέους, ότι πρέπει δηλαδή να επισκευάζουμε τη σκεπή μας όταν έχουμε καλό καιρό και όχι όταν έχουμε κακό καιρό. Τώρα υπάρχουν χώρες με υψηλό χρέος όπως είναι η Πορτογαλία που εποφελήθηκαν από καλούς όρους για την χρηματοδότηση, η επαναχρηματοδότηση του χρέους. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από τον καλό καιρό εντό αγωγικών. Δεύτερον, η τεχνολογία, blockchain ή τα κρυπτονομίσματα, ε, παντός είδους τρόποι ε, πληρωμών Όλα αυτά υπάρχουν. Κάποιος από, το, την Επιτροπή αναφέρθηκε στο Libra, ένα κρυπτονόμισμα ε, που κάποιες εταιρείες σκέφτονται να βάλουν στην αγορά και είπε ότι θα είναι απειλή αυτό. Ποια είναι η καλή ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα του συστήματος και σε κίνητρα για καινοτομία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Απάντηση. Ευχαριστώ. Ναι, να επισκευάζουμε τη σκεπή όταν ε, ο καιρός είναι καλός. Ο Φιτζελ Κέναντι το είχε πει. Όντως, πολλοί χρησιμοποίησαν αυτή τη φράση, πολύ πολιτική και άλλοι. Αλλά πολλοί μείναν στα λόγια και δεν το έκαναν πράξη. Όσο υπάρχει ακόμα ανάπτυξη τώρα, και έχουμε περάσει από μια τεράστια περίοδο ανάπτυξης χωρίς προηγούμενο ε, σε πάρα πολλές χώρες. Και μετά έχουμε απειλές, είτε πρόκειται για το διεθνές εμπόριο, ότι υπάρχει το Brexit, είναι γεωπολιτική κίνδυνη. Για να μην αναφερθώ και στο κλίμα, τα είπαμε αυτά, που είναι πιο μακροχρόνιο θέμα, αλλά απαιτεί άμεσε λύσει. ε, όντως ισχύει αυτό, το ότι πρέπει να επισκευάζουμε τη σκεπή του σπιτιού μα όταν ο καιρό είναι ακόμα καλός. Άλλε χώρες έχουν μεγάλα περιθώρια, άλλες πρέπει να προσαρμόσουν την πολιτική τους και να διευκολύνουν τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Τώρα για το δεύτερο ερώτημά σας που απαιτεί συζήτηση σε βάθος το θέμα των τεχνολογικών αλλαγών και ισορροπία ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος από τέτοιες τεχνολογικές αλλαγές. Η γενική αρχή είναι ότι οι κυβερνήτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να γνωρίζουν τις εξελίξεις, να ενημερώνονται συνεχώς, γιατί οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα καθημερινά και πρέπει να το κάνουν αυτό έχοντας υπόψη στα τα δύο. Πρώτον, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστασία καταναλωτών και επενδυτών. Και δεύτερον, να έχουν υπόψη τους να διευκολύνουν και να επιτρέπουν την καινοτομία. Γιατί οι κεντρικοί τραπεζίτες, όπως και άλλοι πολιτικοί, δεν μπορεί να κλείνουν τα μάτια και να απαριστάνουν σαν να πρόκειται να συνεχιστούν τα πράγματα χωρίς καμία αλλαγή δεν είναι δυνατόν ε, να πηγαίνουν ε, με τον ίδιο τρόπο και να ταξιδεύουν ε, παντού νομίζοντας ότι θα συναντήσουν παντού τις ίδιες συνθήκες. Όχι, η τεχνολογία προχωράει, οι αλλαγές γίνονται. Και το ίδιο ισχύει και για την ΕΚΤ. Ποια από σας ξέρετε τα tips. Ακριβώς αυτό φοβόμουν. Ούτε εγώ ήξερα τι είναι τα tips. Είναι ένα σύστημα που το Νοέμβριο εγκαθίδρυσε η που δεν έχει στεφτεί με μεγάλη επιτυχία ακόμα, όμως έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει απευθείας πληρωμές σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα δούμε αν οι τράπεζες θα το χρησιμοποιήσουν, αλλά είπαμε χρηματοπιστωτική σταθερότητα και καινοτομία. Και να θέτουμε το ερώτημα, πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να είναι εκείνες που βρίσκονται στην αρχή τέτοιων τεχνολογικών επιτεγμάτων όπως τα κρυπτονομίσματα. Πολ Τάγκ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επανέλθω στο θέμα της δημοσιονομικής ικανότητας. Με ενδιαφέρει γιατί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, ήθελε να υπάρχει μια τέτοια, να υπάρχει δημοσιονομική ικανότητα και θέσετε και συγκεκριμένους όρους. Θεωρείτε ότι η καθυστέρηση τη εισαγωγή δημοσιονομική ικανότητα μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τη μακροοικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη πέραν των όρων και προϋποθέσεων που θέσατε. Κάνω αυτή την πολύ συγκεκριμένη ερώτηση σε εσά. Το χρειαζόμαστε ή υπάρχουν κίνδυνοι για την μακροοικονομική σταθερότητα. Ε, δεύτερον, ε, για την Ελλάδα, ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι ο στόχος για το, ε, πλεόνασμα, για το πρωτογενές πλεόνασμα είναι μη ρεαλιστικός και μη βιώσιμος και το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους. Συνεχίζετε να πιστεύετε αυτά τα οποία έχει πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αν ναι, ως πρόεδρος της ΕΚΤ, πώς θα τα χειριστείτε. Τρίτον, χαιρετίζω την έμφαση που θέσατε στη βιωσιμότητα. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και η ΕΚΤ ε, είναι ένα υπόδειγμα και έχει ένα ρόλο να παίξει για την βιώσιμη χρηματοδότηση. Η ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει το γενικό στόχο σύμφωνα με το άρθρο 127 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα ε, για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και το κλίμα. Ε, Θεωρείτε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ο πρωταρχικός στόχος αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει ε, θέσει σε προτεραιότητα τους δευτερογενείς στόχους για την καταπολέμηση του κλίματος. Εσείς θα υποστηρίξετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Απαντώντας πολύ άμεσα, δεν νομίζω ότι αν δεν ε, υλοποιήσουμε αυτόν ε, το μηχανισμό σταθερότητας που εγκρίθηκε αλλά δεν έχει προσδιοριστεί και δεν ε, έχουν οριστεί και συγκεκριμένα ποσά από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών τον Ιούνιο, δεν πρόκειται να κάνει να καταρρεύσει η σταθερότητα της Ευρωζώνης. Παρομοίως, πιστεύω ότι για να ενδυναμωθεί και για να μπορέσει να αποτελέσει πραγματικά νομισματική ζώνη με όλα τα γνωρίσματα μιας νομισματικής ζώνης, θα είναι πολύ χρήσιμο και επιθυμητό να έχουμε αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα, όχι μόνο για λόγους ε, ε, σύγκλησης που είναι επιθυμητό στόχος, αλλά διότι ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοκ και τα προβλήματα, προβλήματα ρευστότητας. η μακροσταθερότητα θα επιβιώσει ακόμη και αν δεν το έχουμε τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το χρειαστούμε στο μέλλον. Για την Ελλάδα και το πρωτογενέ πλεόνασμα είναι μια συζήτηση που συνεχίστηκε με την Τρόικα επί πολύ, ιδίω τα τελευταία χρόνια τη συμμετοχή του Δουνουτού στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι συνεχώ το Δουνουτού έλεγε ότι το 3,5% πρωτογενέ πλεόνασμα, κατά τη γνώμη του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και ακόμη μιλώ ω Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, είναι υπερβολικό στόχο και θέτει υπερβολική πίεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την οποία ελπίζαμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνεχίζει να έχει την άποψη αυτή και βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι σε περίοδο ανάκαμψης ε, και ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επανεξετάσουμε με μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι η δική μου αξιολόγηση. Ε, είναι πολύ χρήσιμο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε ε, το ρόλο της ΕΚΤ σε σχέση με τα προγράμματα, γιατί θυμάμαι τις τεράστιες αυτές συναντήσεις, ατελείωτες συναντήσεις ε, της Ευρωζώνης με άπειρες λεπτομέρειες για το είδος των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Ο Μάριο Ντράγκη και ε, οι υπάλληλοι της ΕΚΤ που ήταν ε, ε, στην αίθουσα συμμετείχαν. Και πραγματικά τίθεται το ερώτημα τι μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ήταν, δεν ήταν η βασική τους αρμοδιότητα. Στο μέλλον η ΕΚΤ θα, θα περιορίζει την εξέτασή της στους τομείς που έχει αρμοδιότητα. Δεν έχουμε πλέον χρόνο, λέει ο Πρόεδρος. Ίσως αργότερα μπορείτε να επανέλθετε. Νταμιάν Καγάμ εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Λαγκάρντ. Περιμένοντας λοιπόν ε, να εφαρμοστεί αυτή η ευρωπαϊκή ταξινομία που αναφέρατε και με βάση και ε, ε, τις κλιματικές εξελίξεις είστε πρόθυμοι να δεσμευτείτε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δημιουργήσετε μια πράσινη μεθοδολογία στο ΕΚΤ για το πρόγραμμα ενεργητικών λαμβάνοντας υπόψη και τις επιχειρήσεις που ρηπαίνουν περισσότερο και αποσύροντας σιγά σιγά τις επενδύσεις ε, της ΕΚΤ ε, από τις ε, επιχειρήσεις που ρηπαίνουν. Το 63% των χρηματοδοτήσεων πηγαίνουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ρηπαίνουν, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Η ΕΚΤ έχει τακτικές συναντήσεις με τους επικεφαλής των μεγάλων τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά δεν έχει μια πλατφόρμα διαρθρωμένου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών θα δεχόσατε να δημιουργηθεί ένα ετήσιο φόρουμ συζητήσεων στο πλαίσιο του οποίου η ΕΚΤ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούσαν να συζητούν την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ως εκπρόσωπος της, όπως μας ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι της Φινλανδική Προεδρίας, ε, δεσμεύεστε να αναθεωρήσετε τους ε, κανόνες ηθικής και διοντολογία της ΕΚΤ για την ε, δημοσιοποίηση των συναντήσεων τη ΕΚΤ με λόμπι και με όλους τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών που σήμερα δεν δημοσιοποιούνται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την τελευταία σας ερώτηση, ξέρω ότι ο κώδικας δεοντολογίας αναθεωρήθηκε εις βάθος μετά από κάποια σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με τους εκπροσώπους ιδιωτικού τομέα. Χαίρομαι που ισχύουν οι σωστοί κανόνες του κώδικα δεοντολογίας και θα ήθελα να εφαρμόζονται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς εφαρμόζονται στην ιεραρχία της ΕΚΤ. Όσο καλύτερα και ε, με όσο μεγαλύτερη διαφάνεια εφαρμόζονται, τόσο καλύτερα για την τήρηση των αρχών της διοντολογίας για να διευκολύνεται και το είδος των επαφών και η ημερήσια διάταξη αυτών των συναντήσεων. Δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή καμία συγκεκριμένη δέσμευση, γιατί ε, ακόμη δεν ε, είμαι επικεφαλής της ΕΚΤ. Τώρα, για ένα ετήσιο φόρουμ. Και πάλι δεν μπορώ να δώσω δεσμεύσεις πρόορες, γιατί δεν βρίσκομαι ακόμη στη θέση της επικεφαλής της ΕΚΤ. Ε, όταν ήμουν στο Δουνουτού, αυτό το οποίο υλοποιήσαμε ε, ήταν πολύ εντατικέ διαβουλεύσεις τέτοιου τύπου. Και ε, όσοι γνωρίζουν τι εργασίε του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου ξέρουν ότι πριν από 10 χρόνια οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών ήταν έξω από το Ταμείο και δημιουργήθηκε ένα επικοδομητικό διάλογο και δεν συμφωνούσαμε ούτε συμφωνούμε πάντοτε απολύτω. Αλλά καταφέραμε μέσω αυτού του επικοδομητικού διαλόγου να βρούμε ε, τρόπο συνεννόησης ε, με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από 189 χώρες ολόκληρου του κόσμου. Στην ετήσια συνέλευση του Δουνουτού, επί τρεις ημέρες γίνεται αυτός ο διάλογος με κατανάλωση ενέργειας και με μεγάλο ενθουσιασμό. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ανταλλαγή εμπειριών και ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών ήταν θεμελιώδους σημασίας για να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσδοκίες της ε, κοινωνίας των πολιτών, για να εξηγήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ποια είναι τα όρια των δράσεών μας και για να μπορέσουμε ε, να προωθήσουμε τις δράσεις μας χάρη στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, Εάν ε, εφαρμόζεται μια ταξινομία η οποία εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να δούμε τη διαδικασία της ε, υλοποίησης αυτής της ταξινομίας και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο ε, εκπομπών άνθρακα και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επενδύσεις για εταιρείε όταν φτάνουν σε περίοδο ορίμανσης οι επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Γκούνερ Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, πιστεύω να ε, οριστείτε στην θέση της ε, Προέδρου της ε, ΕΚΤ. Σας καλωσορίζουμε καταρχήν εδώ. Θέλω να πω το εξή. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν την, τον αναλάβουν όλοι από κοινού δημόσιο χρέος και απαγορεύουν και τη χρηματοδότηση από το κράτος είτε μέσα από εξαγορά ομολόγων είτε μέσα από άλλες κινήσεις. Απαγορεύεται και η αγορά δευτερογενών ε, ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Παρ' όλα αυτά, από το 2010 και κυρίως ε, από τότε που ε, ανέλαβε ο ακόμα πρόεδρος της ΕΚΤ, ο κύριος Ντράγκη, παρ' όλα αυτά, αυτά γίνονται. Ως Γαλλίδα Υπουργός το 2010 και το 2011 είπατε τότε με δική σας πρωτοβουλία και πραγματικά τότε εγώ το είχα εκτιμήσει ιδιαίτερα και το εκτιμώ ακόμα. Είχατε πει λοιπόν ότι κατά την άποψή σας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και η ΕΚΤ έσπασαν, παραβίασαν τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, σώσουν το ευρώ και δεν είσαστε μόνο μία πολύ επιτυχημένη πολιτικός, αλλά και μία ε, νομικός εγνωσμένου κύρους. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, εάν ε, συνεχίσετε, όπως και η προκάτοχή σας, να παραβιάζετε το δίκαιο, παραδείγματος χάρη ε, παρά τη συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκολύνετε και να προβλέπετε ελαφρύνσεις για κράτη και επιχειρήσεις, τότε η σταθερότητα των τιμών κάτι για το οποίο έχετε δεσμευτεί, όπως επίσης και το 2% πληθωρισμός, κατά προσέγγιση 2%, ε, θα μπορούσε, όπως είπατε σήμερα, να ξεπεράσει και το 2%. Ε, κατ' Όλα αυτά τι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι οι καταθέτες, οι φορολογούμενοι και πολλοί άλλοι, οι οποίοι φέρουν τη λιγότερη ευθύνη για την κρίση, αυτοί θα επιβαρυνθούν. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η αρχή της ίδιας ευθύνης στα δημοσιονομικά που και αυτή υπονομεύεται. Και ένα άλλο ερώτημα. Σε τελική ανάλυση, εσείς πώς αιτιολογείτε το δικαίωμα το οποίο διεκδίκησε η ΕΚΤ να είναι πάνω από οποιοδήποτε μορφή δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί ε, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο και υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν το τι είναι νόμιμο και τι καθίσταται παράνομο. Νομίζω μέσα ακριβώς σε αυτά τα όρια πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν οι θεσμοί. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά αρκετές φορές και σε διεθνές και σε περιφερειακό επίπεδο αναγκαστήκαμε να αποκλίνουμε, δεν θα έλεγα απαραίτητα να παραβιάσουμε τις συνθήκες, γιατί υπήρχαν ε, τομείς και θέματα όπου δεν υπήρχαν προβλέψεις, δεν είχε τίποτα προβλεφθεί το τι πρέπει να γίνει για να ε, προστατευτούν παραδείγματο χάρη οι καταθέσεις και οι αποταμιεύσεις των καταθετών. Το 8-9 σχεδόν όλοι είχαν προχωρήσει πέρα από τους κανόνες και αυτό για το κοινό καλό. Γιατί, για να μην χάσουν οι άνθρωποι τις καταθέσεις τους. Ακούω πολύ συχνά αυτούς που μας λένε ότι προστατεύσατε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς απλά διασφαλίσαμε να μην υπάρξει πανικός, τραπεζικός πανικός, ε, να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες για να προστατευτούν οι καταθέσεις. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και δικαιολογημένο και απαραίτητο. Όσον αφορά τώρα το 2% ε, κάτω από αλλά κοντά στο 2% αυτό που συζητιέται στην ΕΚΤ ε, είναι το εξής. Μπορεί να πλησιάσει κανείς το 2% από κάτω, ανεβαίνοντας σιγά σιγά, 1,6, αλλά μπορεί να πάει στο 2% και από πάνω. Και νομίζω ότι αυτό το μεσοσταθμικό το 2% έτσι πρέπει να το ερμηνεύεται. Τουλάχιστον εγώ έτσι κατανοώ και ερμηνεύω τη συζήτηση και είναι σωστό να υπάρχει μια συμφωνία που είναι αποδεκτή και από επάνω αλλά και από κάτω. Επόμενος ομιλητής από το ECR. Χαίρομαι που σας βλέπω, κυρία Λαγκάρτ. Έχω τρεις ε, δηλώσεις και να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που θα πω και αν όχι να μου εξηγήσετε γιατί. Είπατε μόνοι σας προηγουμένως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς ε, τη διαφορά του 1,2% πληθωρισμό ή 1,8% παραδείγματο χάρη ενδεικτικά. Παρόλα αυτά, ε, παρά αυτό το επιχείρημα, το έολο θα έλεγα, ε, υπάρχουν ε, περίεργες πολιτικές ε, που εφαρμόζονται και συνεχίζονται. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Δεύτερον, βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον ε, στο βιομηχανοποιημένο κόσμο ε, τη μείωση της παραγωγικότητας ε, και παραμένουν πολλές φορές εταιρείε ζόμπι όπως αποκαλούνται. Τι είναι αυτές οι εταιρείε, είναι εταιρείε που απλά επιβιώνουν λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων. Με αυτές τις πολιτικές τελικά έχουμε ε, μη αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες αναποτελεσματικές πλήρως και ως εκ τούτου όλες αυτές οι πολιτικές οδηγούν στην ε, χρηματοπιστωτική αστάθεια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις μου. Ευχαριστώ. Μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω αυτό που έλεγα και πριν για το 2%. Δεν είναι για να υποβάσω τη σημασία που έχει αυτή η συζήτηση. Οι παρατηρήσεις ε, είναι πολύ καλές, οδηγούν σε κάποιες προσδοκίες. Η συζήτηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων, δηλαδή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ε, ο Κεντρικός Τραπεζίτης της Αυστραλίας μιλούσε για μια ελάχιστη ευελιξία στην επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό. Συνεχίζει τώρα στα αγγλικά, ενώ πριν μιλούσε γαλλικά η κυρία Λεγκάρ. δεν καταλαβαίνω γιατί μιλούσα γαλλικά και τώρα θα σας μιλήσω αγγλικά για τα υπόλοιπα. Από την άλλη λοιπόν αναφερθήκατε στο θέμα του πολύ χαμηλού κόστος χρηματοδότησης και αυτό διευκολύνει την επιβίωση εταιριών που αν δεν υπήρχε θα είχαν εξαφανιστεί. Ξέρετε και πάλι πρέπει να γίνεται ανάλυση κόστους ωφέλους. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτό το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ε, πόσα θα ήταν τα δάνεια, πόσες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτούσαν τις δαπάνες τους. Υπάρχουν ε, πράγματα της ΕΚΤΟ όπως ο στοχευμένος μηχανισμός χρηματοδότησης και αυτά έχουν στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ε, τώρα μπορούν να βελτιωθούν όλα αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος. Πιστεύω πως πράγματι μπορεί να υπάρξει μία εξειδίκευση. Και τώρα ξεκινάμε ε, στον τελευταίο γύρο των ερωτήσεων. Ε, τέσσερα λεπτά, ο Χωσέ Καρσία Μαγκάλ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, αγαπητή κυρία Λαγκάρτ. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω πάλι εδώ. Έρχεστε σε κάποια στιγμή διαφορετική από εκείνη που έφτασε ο κύριος Δράγκη το 2015 εν μέσω μιας υπαρξιακής κρίσης, με περιθώρια λιγμών όμως στην ομισματική πολιτική μέσω των επιτοκίων κλπ. Εσείς ε, φτάνετε όταν ο ήλιος μεν λάμπει, αλλά που υπάρχουν σύννεφα μαύρα στον ορίζοντα. Και όταν η νομισματική πολιτική έχει ήδη επιτόκια πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, ποια θα είναι η φύση της νέας κρίσης, θα είναι διαφορετική. Δεν θα είναι κρίση ζήτησης, αλλά κρίση προσφοράς από ό,τι φαίνεται. Οπότε ο ρόλος των διάφορων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας θα είναι διαφορετικός. Βραχυπρόθεσμα, όντω μπορούμε να παίξουμε με τη δημοσιονομική και την νομισματική πολιτική, αλλά πιο μακροπρόθεσμα χρειάζεται να έχουμε μεταρρυθμίσει. Σας ρωτώ λοιπόν το εξή. Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία, για να μην μιλήσουμε για την παγκόσμια, μπορεί να συνεχίσει με αρνητικά επιτόκια χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα του συστήματος και τράπεζες. Δεύτερον, λαμβάνοντα υπόψη το ρόλο που θα παίξουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενεργητικού, ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε τον κανόνα που συνδέει την αγορά χρέους μιας χώρας ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας του και να αλλάξει και να υποφεληθούν οι χώρες οι οποίες χρωστούν. Έπειτα, η εμπειρία δείχνει ότι υπήρξε κάποια προτίμηση για τα κρατικά ομόλογα. Μήπως θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο στα, στο εταιρικό ενεργητικό. Μήπως θα ήταν λογικό το καλάθι των ενεργητικών που επιλέγονται να μεγαλώσει και να μην περιοριστούμε μόνο ε, στο τραπεζικό. Ευχαριστώ πολύ και Επαναλαμβάνω και πάλι, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, ελπίζοντας ότι θα αναλάβετε τα καθήκοντά σας επικεφαλής της ε, ΕΚΤ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας δω και σε άλλες ε, συνθήκες. Λοιπόν, με ρωτάτε κάτι πολύ συγκεκριμένο, χωρίς να μπορώ εγώ να δώσω πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Πόσο καιρό θα έχουμε ακόμα αρνητικά επιτόκια? Μα δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Γιατί η σταθερότητα τιμών είναι το καθοριστικό. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν χρησιμοποιούνται πλήρως. Και ακόμα υπάρχει περιθώριο για να αναπτύξουμε κάποια από αυτά περισσότερο. Οπότε είναι δύνατο να πω τώρα πότε και κάτω από ποιες συνθήκες και πώς. Γιατί πρέπει να γίνει πρώτα μια ανάλυση κόστους-οφέλους ε, της χρήσης των μέσων αυτών. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας, και είναι νομίζω, ότι το πρόγραμμα αγοράς θα παραμείνει ως έχει μέχρι να μην ε, ανέβουν τα επιτόκια. Ξέρω δηλαδή ποια σειρά θα ακολουθήσουμε. Οπότε αυτό βλέπουμε προς το παρόν. Τώρα, δεν ξέρω τι εννοείται μιλώντας για αγορά ομολόγων από τις εντό καλές ή λιγότερο καλές χώρες. Ε, δεν ξέρω αν εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε την ηθική μέσα σε αυτήν την άσκηση αντοχής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα κλειδιά της ΕΚΤ για να μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει με τις αγορές αυτές. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει. Τέλο πάντων, μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως αργότερα μεταξύ μας. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι αναφέρεστε στο σύστημα tiering, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Ωραία. Εργίν Ερόγλου από το Renew. Παρακαλώ. Α, δεν είναι. Α, είναι εκεί, είναι. Αξιότιμη κυρία Λαγκάρτ, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Ε, τις τελευταίες δύο ώρες ε, τέθησαν αρκετά ερωτήματα, γι' αυτό ε, θέλω να εμβαθύνω κάτι, το θέμα των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών νομισμάτων. Τα τελευταία χρόνια αυτά διαδίδονται όλο και περισσότερο και θέλω να ρωτήσω, αυτά αποτελούν ανταγωνισμό, ανταγωνιστικά νομίσματα στο ευρώ. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η εγκληματική και κατά πόσο είναι καθήκον της ΕΚΤ να αναχαιτήσει αυτή την εξέλιξη. Ε, ίσως ε, να δίδει και κάποιες συμβουλές ε, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και κάτι άλλο που δεν ετέθη σήμερα εδώ. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή η πολιτική της ΕΚΤ με τα αρνητικά επιτόκια αντιμετωπίζεται πολύ επικριτικά γιατί αυτή η πολιτική κυρίως ε, για τα μικρά ταμιευτήρια στη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα. Κατά την άποψή σας ε, είναι απαραίτητο να υπάρξει συρρήκνωση του αριθμού των ε, τραπεζικών ιδρυμάτων ή θα μπορούσε στη Γερμανία να εκτιμήσει κανείς ότι με αυτή την πολιτική ενδεχομένως υπάρχουν ενδείξεις για μια επερχόμενη κρίση. Θα ήθελα ή δυνατόν να, μας, ε, να μου απαντήσετε. Φαντάζομαι δεν με ρωτάτε τι πιστεύω για μια συγκεκριμένη συγχώνευση τραπεζικών ιδρυμάτων. Λοιπόν, πάμε πίσω ε, στα ψηφιακά νομίσματα, ε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή καταρχήν ε, χρηματοπιστική σταθερότητα και αποφυγή και αποφυγή προβλημάτων. Ξέρετε, εγώ ε, θα ήθελα να διαφοροποιήσω τα διάφορα κρυπτονομίσματα που βεβαίως ε, αυτά αναλύονται διαφορετικά ανάλογα με το που ακριβώς ε, αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν χώρες όπου αυτά τα νομίσματα αντιμετωπίζονται ως κεφάλαιο, ως ασφάλεια. Υπάρχει δηλαδή ένα ολόκληρο χάος για το σωστό πλαίσιο. Αλλά εντωμεταξύ έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ε, ιδιαίτερα μεταβλητό προϊόν, το οποίο όμως δεν απειλεί την σταθερότητα, δεν είναι εμπόδιο για την σωστή εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Εγώ αυτό θα το διαχώριζα από τα σταθερά νομίσματα, που κατά την άποψή μου είναι κάτι τελείως διαφορετικό και που ε, έχουν και διαφορετικό μέλλον. Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι τα σταθερά νομίσματα, είτε είναι λίμπρα είτε οτιδήποτε άλλο, η κεντρική τράπεζα ως προς τα ψηφιακά νομίσματα, αυτά τα ψηφιακά νομίσματα θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς. Δεν με απασχολεί τόσο κατά πόσον πρόκειται για τράπεζα ή όχι. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η δραστηριότητα που αναπτύσσεται έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η συμμόρφωση με τους ε, κανόνες. Και γι' αυτό το λόγο εγώ θα έλεγα ότι οτιδήποτε μας προστατεύει από την ομοιοποίηση παράνομων εσόδων, από τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας, από τη σωστή εφαρμογή των νομισματικών πολιτικών, όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οποτεδήποτε επιτραπεί να κυκλοφορούν αυτά τα νομίσματα εδώ αλλά και σε άλλες περιοχές. Γιατί χάρηκα όταν άκουσα ότι η ΕΚΤΕ εκλήθη από το G7 να εξετάσει τα ψηφιακά νομίσματα και να υποβάλει το στομό των δυνατών τα πορίσματά της. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Λαγκάρτ εγώ θέλω να σας πω, πριν από κάποιους μήνες ήμουν παρόν στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, μπροστά σε όλους τους ε, πολιτικούς ε, ομολόγησε ότι άκουσε υπερβολικά τις απόψεις ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και έτσι εφαρμόστηκαν πολιτικές λιτότητες που μεταξύ άλλων γονάτισαν και τον ελληνικό λαό. Και σας ερωτώ, εφόσον ήταν σαφές ότι η κρίση του 2008 οφείλεται σε έλλειψη ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, η οι οικονομολόγοι, οι θεωρητικοί, πολλοί από αυτούς αναφέρετε κι εσείς, εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι οι αγορές πρέπει να αυτορυθμίζονται. Και οι δυσλειτουργίες που υπάρχουν η ανισότητα για την οποία μιλήσατε προηγουμένως, αυτά οφείλονται ε, κυρίως ε, σε κακές πολιτικές και όχι στην έλλειψη των ρυθμίσεων. Εσείς μιλήσατε ότι δεν εφαρμόζονται οι συνθήκες και εγώ σας ερωτώ, ποια είναι η δική σας η άποψη ως προς το ενδεχόμενο το να αναθωρηθούν οι συνθήκες, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει μια νέα λειτουργία, δηλαδή να είναι... Ε, το τελευταίο καταφύγιο για τις ε, διάφορες χώρες ανάλογα με τις ανάγκες τους και ως εκ τούτου στο καταστατικό ε, της ε, τράπεζας να είναι πρώτα απ' όλα η αντιμετώπιση της ανεργίας και όχι τόσο η σταθερότητα των τιμών. Well, any Οποιαδήποτε αλλαγή την εντολή της ΕΚΤ ε, εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εφεύρει η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τη σταθερότητα των τιμών σε σταθερότητα των τιμών συν καταπολέμηση της ενεργείας, συν βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει στο άρθρο 127 υποπαράγραφος 2 ένα σημείο το οποίο επιτρέπει στην ΕΚΤ ε, παράλληλα με την ε, ικανοποίηση του πρωταρχικού στόχου της σταθερότητα των τιμών να εξετάζει και του δεύτερογενεί στόχου που τίθενται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να διευκρινίσω και κάτι για μια προηγούμενη ερώτηση, ότι το περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος, αν θυμάμαι σωστά, είναι τμήμα αυτών των στόχων. Αυτό, επομένως, νομιμοποιεί την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως δευτερογενούς στόχους που έχει πρωταρχική σημασία αλλά αποτελεί ένα δευτερογενή στόχο του, ε, της ΕΚΤ. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας για το ποιος έκανε τι σε σχέση με ε, τα μνημόνια στην Ελλάδα. Πάντω και εδώ το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ιδίω στο τελευταίο τμήμα των προγραμμάτων, ε, έχει καταγραφεί ότι δήλωσε ότι οι απαιτήσει έναντι τη Ελλάδο ήταν υπερβολικέ σε σχέση με τι δυνατότητε τη και ότι το πρωτογενέ πλεόνασμα του 3,5% πρέπει να εγκαταληφθεί προ κάτι περισσότερο γραμμικό και πιο κοντά στο 1,5 έω 2% κατά μέγιστο. Ε, κοιτάξτε, υπήρχε η Τρόικα λαμβάνονταν πολλές αποφάσεις από πολλούς φορείς. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αρχίσουμε να κατηγορούμε τον έναν ή τον άλλον. Ήταν μια κοινή προσπάθεια. Και αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Η Ελλάδα μας είχε ζητήσει τη βοήθειά μας. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή, αλλά είναι αλήθεια ότι υπέφερε λόγω του προγράμματος αναδιάρθρωσης που εφαρμόστηκε. Ευχαριστώ. Η Ρένε την άλλη από τους σοσιαλδημοκράτες. I can, but maybe not everybody. Το μικρόφωνο δεν είναι ανοιχτό. Okay. Thank you. So, a lot is... Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχει συζητηθεί πολύ το θέμα των πράσινων ομολόγων. Πολλά από τα προηγούμενα ερωτήματα αφορούσαν την πλευρά της ζήτησης. Όπως σωστά είπατε και στην απάντησή σας στις ερωτήσεις, ε, έχουμε πρόβλημα ε, προσφοράς. Και στο ερώτημα αυτό ανοίγεται και τη δυνατότητα δημόσιας παρέμβασης για να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο περιβάλλον για αυτή την αγορά. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Θα ήσασταν υπέρ ε, μιας μεγάλης δημόσιας έκδοσης πράσινων χρηματοπιστωτικών εργαλείων από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζετε ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτή την έκδοση, όχι αγοράζοντας την ιδιωτική αγορά που δεν ε, επιτρέπεται από τη συνθήκη, αλλά να τα δέχεται ε, ως εγγυήσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά τα ομόλογα σε σχέση με άλλους τύπους ομολόγων. Δεύτερο ερώτημα, τα κρυπτονομίσματα. Είπατε ότι δεν αποτελεί, αποτελούν απειλή στο, στα παραδοσιακά νομίσματα ή στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το καλοκαίρι ακούστηκε η στην χρηματοπιστωτικη σταθεροτητα το καλοκαιρι ακουστηκε η ιδεα των κρυπτονομισμάτων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα αντίβαρο στην ηγεμονία του δολαρίου. Θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σας σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις και τι απαντήσεις θα μπορούσε να δώσει η ΕΚΤ σε αυτό. Ευχαριστώ. Για την πρώτη σας ερώτηση για τα πράσινα ομόλογα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή, Επενδυτική η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, είναι εκδότης τέτοιων ομολόγων και η ΕΚΤ στην ε, δευτερεύουσα αγορά αγοράζει κάποια τέτοια προϊόντα και το κατόφλι μέχρι το οποίο μπορεί ε, να έχει τέτοια ομόλογα δεν είναι 33% αλλά 50% άρα τις επιτρέπεται να έχει ε, περισσότερα ε, βράσινα ομόλογα σε σχέση με άλλα ομόλογα και αυτό είναι θετικό. Επίσης χαίρομαι διότι η Ursula von der Leyen προωθεί ενεργά μια νέα πράσινη συμφωνία. Είναι της γνώμης ότι η έκδοση αυτών των ομολόγων έχει κέρια σημασία και συμφωνώ απολύτως. Για τα κρυπτονομίσματα, και για την πρόταση του Μακάνη. Με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ. Μου κίνησε το ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Δεδομένων των συνεχών εξελίξεων. Με δύο λόγια να πω για αυτούς που δεν διάβασαν την ομιλία του Μακάνη, αυτό που προτείνει είναι κάποιες από τις βασικές κεντρικές τράπεζες να σχηματίσουν μια κοινοπραξία και να διερευνήσουν κατά πόσο είναι δυνατόν να δημιουργήσουν νομίσματα των κεντρικών τραπεζών, κοινά νομίσματα. Αυτό που έχει κατά νου το Λίμπρα δηλαδή, αυτοί που επινόησαν το Λίμπρα, να υπάρχει ένα εργαλείο μετατρέψιμο ε, σε ε, κρατικά νομίσματα. Ο Μακάνη προτείνει κάτι παρόμοιο, αλλά θα είναι κάτι το, θα το οποίο θα εκδίδουν οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες. Και όντως ε, αυτό έχει αρκετές ενδιαφέρουσες πτυχές. Μπορούμε να τις διερευνήσουμε. Δεν μπορώ να προδικάσω ποια θα είναι η άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αλλά προσωπικά θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διερεύνηση αυτής της νέας έννοιας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ εκπροσωπώ τους πολίτες μιας χώρας που δεν είναι στην Ευρωζώνη, την Ουγγαρία. Και θέλω να σε ρωτήσω το Πρώτον, για τη συνεργασία μεταξύ χωρών Ευρωζώνης, χώρες χωρίς της Ευρωζώνης. Είναι ζωτική σημασία να υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών χωρών. Ό,τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη επηρεάζει πάρα πολύ τις χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Ε, είναι αυτό που λέμε ότι βύχης ε, στην Ευρωζώνη παθαίνει πνευμονία ε, κάποιος που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Οπότε θέλω να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει μια νέα πρόταση η οποία εγκρίθηκε εν μέρη για την δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης και σίγουρα το γνωρίζετε ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές ανησυχίες στις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Στη γραπτή σας απάντηση είπατε ότι σας, σας ικανοποιεί μια τέτοια πρόταση. Οπότε πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες αυτές που εκφράζουν οι χώρες που δεν είναι στο ευρώ, που δεν έχουν το ευρώ. Και τι γίνεται με τις προϋποθέσεις ένταξης στην Ευρωζώνη. Γιατί υπάρχουν ότι προηγουμένως πρέπει να συμμετέχουν σε δομές κτλ. Οπότε θέλω να ρωτήσω, οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα είναι επαρκής ή νομίζετε ότι θα δημιουργήσετε και άλλες προϋποθέσεις. Γιατί έτσι θα ξέρουμε και εμείς αν απεξερχόμαστε επαρκώς στις υποχρεώσεις μας και είμαστε έτοιμοι ή όχι να μπούμε. Τέλος, για τα μαθήματα που έχουμε πάρει από την τελευταία κρίση, η χώρα μας χρησιμοποίησε η Ουγγαρία ε, μεικτά μέσα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ε, πολλά από αυτά βέβαια δεν άρεσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φαίνεται ότι λειτουργήσαν. Γιατί για δεύτερη χρονιά η Ουγγαρία έχει την μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Ήδη εσείς είπατε ότι ήταν πολύ καλή δράση της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά και οι χώρες μέλη για να αποφύγουν μια νέα απειλή, μια νέα κρίση. Τι θα πρέπει να γίνει διαφορετικά τώρα από τις χώρες μέλη για να αποφευχθεί μια πολύ χαμηλότερη ανάκαμψη στην Ευρωζώνη σε σχέση με αλλού. Απάντηση. Η συνεργασία ανάμεσα στις χώρες Ευρωζώνης και μη Ευρωζώνης είναι πάρα πολύ σημαντική, το πιστεύω και εγώ αυτό. η επιθυμία είναι να είναι 26 εκτός από τις χώρες opt-out, Δανία και ελπίζουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να λύσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο το θέμα του. Η συνεργασία λοιπόν είναι ζωτική σημασία γιατί είμαστε όλοι μέλη τη ίδια οικογένεια. Θα ζούμε μαζί. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική πράγματι. Ναι, όντω. Καλωσόρισα την ενδρυγική μορφή της δημοσιονομικής ικανότητας που αναφέρθηκε τον Ιούλιο ε, και την ε, καλωσορίζω, τη βλέπω θετικά σαν ένα πρώτο βήμα, γιατί μπορεί να βοηθήσει στη σύγκληση κλπ. Αλλά ίσως να πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά, εφόσον οι προϋποθέσεις το επιτρέπουν και οι χώρες μπορούν να ακολουθήσουν. Και πάλι λοιπόν η συνεργασία με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης είναι σημαντική, γιατί κάποια στιγμή θα μπουν σε αυτή την ομάδα. Ελπίζω να προχωρήσουμε κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις. Επιπλέον προϋποθέσεις ε, για να μπορούν να ενταχθούν ε, οι χώρες στο ευρώ. Το είδαμε και στην περίπτωση της Κροατίας ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Μπαίνουν στην ε, Τραπεζική Ένωση, τηρούν τις αρχές, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Εγώ προσωπικά Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος στο θέμα της καταπολέμησης νομιμοποίησης ε, χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες και αντιμετώπιση και καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών. Δεν λέω ότι αυτά που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας αρκούν. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και σίγουρα βοηθάει η συνεργασία. Ο κ. Παπαδημούλης, παρακαλώ. Ε, σας καλωσορίζω κυρία Λαγκάρτ. Σημειώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση όσα είπατε για την ανάγκη να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια για τη χώρα μου. Και σημειώνω επίσης με ικανοποίηση την επισήμανσή σας ότι η ελληνική οικονομία σημειώνει μια ισχυρή ανάκαμψη το τελευταίο διάστημα, πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Πριν λίγο δόθηκαν τα επίσημα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, με μια ανάπτυξη 1,9%. Ελπίζω την πρότασή σας να την ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργό, ο νέος Έλληνας Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκη, έτσι ώστε να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η χώρα μου, ε, συζητώντας με τους δανειστές, για πιο χαμηλά ρεαλιστικά πλεονάσματα. Ελπίζω να είναι το ίδιο φιλόδοξος με εσά σε αυτή τη διεκδίκηση. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, όμως και για όσα υπέφερε η χώρα μου και ο λαός μου, ιδιαίτερα στα πρώτα δύο μνημόνια. Ο κύριος Ντομινίκ Ροσκάν, ο κύριος Ντάισεμπλουμ, μίλησαν για τους περίφημους λάθος πολλαπλασιαστές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που προκάλεσαν τριπλάσια ανεργία, και μια ύφεση διπλάσια αυτών που υπολογίζατε ως Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είπαν με θάρρος ότι αυτά έγιναν, όπως και η μία αναδιάρθρωση του χρέους, για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των γαλλικών και γερμανικών τραπεζών. Εσείς ποια γνώμη έχετε, γιατί οι δύο κύριοι που ανέφερα είναι τέος πλέον. Εσείς εφαρμόζετε ένα παράδειγμα ανακύκλωσης. Περνάτε από την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα είχε λοιπόν σημασία να μας πείτε τη γνώμη σας, γιατί το κουτί της Πανδώρας άνοιξε πριν από πολλά χρόνια σε βάρος της χώρας μου και δεν θα ανοίξει τώρα αν είμαστε όλοι ειλικρινείς. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να έχει περισσότερη διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία από το Ευρω... Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για να ενισχύσετε αυτή τη διαφάνεια. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαδημούλη. Νομίζω ότι αυτά που είχα να πω για το πρωτογενές πλεόνασμα στην Ελλάδα τα είπα. Και είπα επίσης ε, το πόσο αγωνιστήκαμε για να περάσουμε τη δική μας τη θέση. Τη δική μου τη θέση που ήταν διαφορετική. Ε, γι' αυτό το λόγο ε, δεν θελήσαμε να αλλάξουμε στην τρίτη φάση του προγράμματος. Πράγματι, είναι αλήθεια, πολλές από τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές ήταν ένα κομμάτι του συνολικού πακέτου και εκεί ε, δεν υπήρξε ε, σωστή εφαρμογή. Θέλω να ελπίζω ότι η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα θα συνεχίσει αυτά που έχουν ήδη ξεκινήσει, θα εμβαθύνει όμως περισσότερο, ε, θα καταστήσει την ε, Ελλάδα ανταγωνιστικότερη. Εγώ χαίρομαι που υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και χαίρομαι ε, που στην Ελλάδα πλέον ξεκινάνε περισσότερες τουριστικές αλλά και μεταποιητικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τον δημοσιονομικό συντελεστή, τον πολλαπλασιαστή μάλλον, το αναγνωρίσαμε αυτό, όχι μόνο σε σχέση με εσά, αλλά και σε σχέση με την Πορτογαλία. Τότε που εξετάσαμε τι επιπτώσει του πολλαπλασιαστή στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Αναγνωρίσαμε ότι είχαμε υποεκτιμήσει, υποτιμήσει ε, τι επιπτώσει από τον πολλαπλασιαστή και γι' αυτό θελήσαμε να αναπροσαρμόσουμε τα μέτρα ε, που θα έπρεπε να ληφθούν ε, βάσει του προγράμματος. Πράγματι, δεν ήταν όμως ευθύνη ενός μόνο ή δύο οργανισμών, όλοι έφεραν κατά κάποιον τρόπο την ευθύνη και γι' αυτό δεν έχει νόημα τώρα να αποδίδει κανείς ε, υπετιότητες. Είναι βέβαια σημαντικό να αναγνωρίζει κανείς όταν κάτι δεν είναι σωστά σχεδιασμένο ε, να το αναγνωρίζει και νομίζω ότι εμείς ε, το κάναμε με απόλυτη σαφήνεια. Εμείς έχουμε ένα εσωτερικό μηχανισμό, έχουμε ένα γραφείο που κάνει εσωτερικές αξιολογήσεις και εκεί λοιπόν έχει συζητηθεί επανειλημμένα το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα στη διαφάνεια, εγώ είμαι στο να υπάρχει ως το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια που να είναι και συμβατή με την ανεξαρτησία του θεσμού. Ε, όμως θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι η συζήτηση που θα γίνει, αν τελικά οριστώ, διοριστώ, ε, τέσσερις φορές το χρόνο, πέντε φορές με την Επιτροπή και μία φορά στην Ολομέλεια, όλα αυτά θα είναι ένα κομμάτι της διαφάνειας υπέρ της οποίας ε, τάσσομαι ανεπιφύλακτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε άλλες πέντε ερωτήσεις. Ε, και άλλες δύο ερωτήσεις στο Κάτσι. Αν δεν τελειώσουμε στη μία, θα συνεχίσουμε μετά τη μία στα αγγλικά. Για να μπορέσετε κι εσείς, ε, κύριε Λαγκάρτ, να ε, κάνετε την καταληκτική σας ε, παρέμβαση. Ίσως μπορούμε να τελειώσουμε μία και πέντε. Αν είσαστε αρκετά γρήγοροι και αν είσαστε και πιο στοχευμένοι. Γιώαχήμ Σούστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν τεθεί πάρα πολλέ ερωτήσει, γι' αυτό και εγώ θα περιστώ σε δύο μόνο θέματα. Αφενό, ε, για μένα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική των χαμηλών επιτοκίων τη στιγμή που πάρα πολλά κράτη εφαρμόζουν μια περιοριστική ε, δημοσιονομική πολιτική. Βέβαια, αυτή η πολιτική τη ε, Κεντρική Τράπεζα έχει και αρνητικέ επιπτώσει, παρέμοντο χάνει στα αρνητικά επιτόκια. Τώρα στη Γερμανία ε, έγινε μια πρόταση από ένα συγκεκριμένο κόμμα όπου λένε από τον νόμο να απαγορεύεται οι τράπεζες ε, να εξακολουθούν να εφαρμόζουν αρνητικά επιτόκια σε καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Εσείς αυτό το βρίσκετε σωστό ή τι έχετε να μας πείτε. Κατόπιν, όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων στην Ευρωζώνη, το αποτέλεσμα των συζητήσεων είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια σε διάφορα κράτη. Αυτό όμως είναι ανόητο, διότι έχουμε κράτη με υψηλότερο δανεισμό και με τον τρόπο αυτό έχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα οι χώρες αυτές να αποπληρώσουν τα χρέη τους και μόνο αυτό, αλλά αποδυναμώνεται και το ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ στο πλαίσιο του να υπάρχει ένας ενιαίος νομισματικός χώρος και μια ενιαία κοινή αγορά, ε, δεν είναι αυταπάτη το να θέλει κανείς να αποφύγει την κοινή διαχείριση κινδύνων. Και μία ερώτηση, τι μέτρα θέλετε να λάβετε έτσι ώστε στην Ευρωζώνη υπάρχει πραγματικά μία δίκαιη διαχείριση κινδύνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνδέετε τα επιτόκια και την δημοσιονομική πολιτική που πρέπει να εφαρμόσουν κάποια κράτη-μέλη. Νομίζω ότι όλα εντάσσονται στην ίδια συζήτηση και όλα αυτά εκφράζουν και αυτά που ε, λένε κεντρικοί τραπεζίτες, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, διάλογος έτσι ώστε ε, να μπορεί να μετρηθεί το κόστος και το όφελος μέτρων τα οποία είναι απαραίτητα έτσι ώστε να φτάσει κανείς και στην επιθυμούμενη σταθερότητα τιμών. Επίσης πιστεύω ότι κάποια μακροπροληπτικά μέτρα ε, πρέπει να εφαρμόζονται για να αντιμετωπίζονται κίνδυνοι σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτά πρέπει να συνεχίσουν ε, και πρέπει ε, να εφαρμόζονται όταν υπάρχει αστάθεια. Πρέπει να σας πω, ανησυχώ ιδιαίτερα σχετικά με το θέμα της ε, μόχλευσης των ε, δανείων. Ε, προφανώς πολλοί τραπεζίτες εστιάζουν σε αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να το ελέγχουμε πολύ προσεκτικά για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την διαμόρφωση κινδύνων. Υπάρχουν τα κάποια μακροπροληπτικά εργαλεία, αλλά θα πρέπει και αυτά να ε, χρησιμοποιούνται σωστά. Καλύτερη διαχείριση κινδύνων στην ε, Ευρωζώνη, αυτό είναι ο τελικό στόχο. Διότι η νομισματική ένωση θα πρέπει να αφορά ε, τόσο του κινδύνου, όσο και την κοινή διαχείριση της ε, επιβράβευσης αν θέλετε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα βέβαια σε αυτό το σημείο. Η Ευρωζώνη ακόμα δεν έχει εκπληρώσει όλους τους, τους στόχους. Υπάρχουν ακόμα κάποια που υπολείπονται. Αν δείτε λιγάκι το θέμα των απολόγων σε διάφορες, κάθε μία χώρα, βλέπουμε ότι ε, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην απόδοση και είναι εντυπωσιακό το πώς ε, τα τελευταία τρίμηνα υπήρξε και μία σύσφυξη. Τώρα, είναι αυτός ο δρόμος προς ε, ένα ελάχιστο spread που είναι αποδεκτό για να υπάρχει διαχείριση και εξάπλωση κινδύνων. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και όπως ανέφερε σήμερα το πρωί ο κύριος Ενρία να ολοκληρωθεί το θέμα των κόκκινων δανείων, αυτά που συνεπάγονται στους ισολογισμούς. Πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά πριν ακόμα περάσουμε στην κοινή διαχείριση κινδύνων, κάτι στο οποίο αναφερθήκατε και που θα ήταν ιδανικό αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Πρέπει όμως να δουλέψουμε πάνω στις προϋποθέσεις για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να μετακινηθούμε στη σωστή κατεύθυνση. Uh, Κύριο από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαγκάρντ. Ίσως αποφύγαμε τα χειρότερα, δηλαδή να μπουν επικεφαλής της ΕΚΤ ε, ε, αυτούς που είναι λαϊκιστές. Με το οικονομικό σενάριο που έχουμε τώρα, θα χρησιμοποιηθεί η εργαλειοθήκη που μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στο παρελθόν. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά τις παρενέργειες αυτών των πολιτικών που πρέπει να εξεταστούν. Σε προηγούμενη απάντησή σας ε, αναφέρατε ε, τις ε, επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων. Έχουν αυξηθεί οι τιμές των ακινήτων και είναι πραγματικό πρόβλημα για τις πόλεις μας η πολιτική της μη αύξηση των επιτοκίων είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά θα πρέπει και να αντισταθμίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Τι να κάνουμε με τα μακροπροληπτικά ρυθμιστικά εργαλεία, όπως είπατε πριν. Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τα αντικυκλικά προστατευτικά μέτρα ε, και άλλες εγγύησεις για να αντισταθμίσετε τα αρνητικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Για το συγκεκριμένο αυτό τομέα, τα ε, μακροπροληπτικά εργαλεία τα οποία πρόσφατα χρησιμοποιήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους για την αγορά κινήτων. Αν δείτε πώς επηρεάστηκε η αγορά κινήτων στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε διάφορες χώρες όπως αυτές, όπου υπήρχε μια έκρηξη των τιμών στην αγορά κινήτων, τα εργαλεία μακροπροληπτικά, είτε είναι δείκτης δανείων προς εισόδημα, είτε κάτι άλλο, ήταν αποτελεσματικά και πρέπει να χρησιμοποιούνται. Στις παρούσες συνθήκες νομίζω ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται. Και να προσθέσω πολύ σύντομα ότι πιστεύω ότι είναι και θέμα προσφοράς. θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών και ίσως να μπορεί να διευκολυνθεί αυτός ο τομέας, ίσως και με δημόσιες επενδύσεις. Αντώνιο Ρινάλντι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λαγκάρντ. διεξάγεται μια συζήτηση σε σχέση με την έντολη της ΕΚΤ και σε σχέση με τις δημοσιοποιήσεις στοιχείων. Και απαντήσατε και σε προηγούμενη ερώτηση συναδέλφου. Είπατε ότι ο πρωτογενής στόχος της ΕΚΤ είναι η σταθερότητα των τιμών και η αποφυγή του πληθωρισμού. Αλλά και πολλοί εθνικοί φορείς θεωρούν την απασχόληση ως πρωταρχικό στόχο. ίσως ο στόχος της ε, απασχόλησης να μπορέσει να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο. Αυτή την ερώτηση θέλω να σας θέσω, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή τη χρονική στιγμή. Ένα δεύτερο ερώτημα. Μπορείτε αυτή τη χρονική στιγμή να εγγυηθείτε στους πολίτες της Ευρώπης την απόλυτη ανεξαρτησία σας. Και αυτό το ερωτώ ως απλός πολίτης της Ευρώπης. Τον Ιούνιο του 2013, όταν δημοσιεύτηκε αυτή η επιστολή στη Λεμόντ, είπατε ότι δεν θέλουμε καν να τα ακούσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αν εγώ γίνω ε, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, ε, τότε είπατε στον κύριο Σαρκοζή, χωρίς ε, την ε, κατεύθυνση θα είμαστε αναποτελεσματικοί, δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Έχουμε ανάγκη έναν άνθρωπο στην αρχή της ΕΚΤ που να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστος και ανεξάρτητος. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να μας διαβεβαιώσετε ότι εσείς σε αυτή τη θέση θα είσαστε απόλυτα ανεξάρτητοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Γιατί νομίζω για το θέμα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας ε, και για το θέμα της ανεξαρτησίας ε, του Προέδρου της ΕΚΤ, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι ναι, πιστεύω ότι συνδέεται εν με την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της Κεντρικής Τράπεζας πολιτικά περιβάλλοντα, αν ανήκει κανείς στο γραφείο ενός υπουργού, αν ε, λειτουργεί μόνος του και δεν έχει την υποστήριξη του ηγέτη, δεν έχει επαρκή αξιοπιστία. Στην περίπτωση του Προέδρου της ΕΚΤ, αυτό το βλέπω ως εντελώς διαφορετική, διαφορετική περίσταση και είναι κάτι ε, το οποίο το παρέχει και ο νόμος. Ε, ο νόμος ζητάει από τους ηγέτες των κρατών μελών να μην ασκούν πίεση στον επικεφαλής της ΕΚΤ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα θεσμικό όργανο που υπηρετεί τους πολίτες της Ευρωζώνης και όχι τους ηγέτες των κρατών μελών και λογοδετεί στους πολίτες της Ευρωζώνης μέσω ημών που είστε οι εκπρόσωποι των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κατά με λοιπόν είναι κέρια σημασία αυτό και χωρίς αυτή την ανεξαρτησία δεν θα είχα καν σκεφτεί να υποβάλω υποψηφιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Στη διαδικασία του Catch the Eye, δύο ερωτήσεις. Ε, θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ε, παρέμβασή σας. Χαίρομαι για την υποψηφιότητά σας για την Προεδρία της ΕΚΤ η αξιοπιστία που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι και γιατί είστε και η πρώτη γυναίκα υποψήφια. Σήμερα είμαστε πέντε γυναίκες από τους 24 ομιλητές που έλαβαν το λόγο. Καμιά φορά η ποιότητα υπερισχύει της ποσότητας. Μου κάνει το πολλό το F. Εγώ είμαι από την Νορμανδία, νομίζω όπως και εσείς κύριε Λαγκάρντ. Και νομίζω ότι οι μεγάλες ε, ε, αλλαγές για το κλίμα, για την τεχνολογία και για άλλα θέματα, μας υποχρεώνουν να επανεξετάσουμε την οικονομική και νομισματοπιστωτική στρατηγική μας. Το ερωτηματολόγιο ε, με τις απαντήσεις σας δείχνετε ότι ε, σκέφτεστε ε, την επανεξέταση της θέσης της ΕΚΤ έναντι των πολιτών, ώστε να ακούτε περισσότερο τη γνώμη των νέων και της κοινωνίας των πολιτών στην ε, Επιτροπή μας ε, θέλουμε μια νομισματική πολιτική που να ε, υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα συμφέροντα των καταναλωτών, γιατί οι καταναλωτές είναι οι βασικοί οικονομικοί παράγοντες. Για όλα αυτά λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε τη δράση της ΕΚΤ περισσότερο κατανοητή, περισσότερο συγκεκριμένη και περισσότερο ανοιχτή παραδείγματος χάρη μέσω των ετησίων φόρουμ που πρότεινε κάποιος συνάδελφος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Χαιρετίζω την Αντιπρόεδρο και ως γυναίκα και ως ε, καταγόμενη από την Ορμανδία, όπως είπατε. Τα ετήσια φόρουμ που αναφέρθηκαν είναι όντως ένας τρόπος να συμπεριλάβουμε την κοινωνία των πολιτών, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί αυτό. Και πιστεύω συγκεκριμένα ότι για να μπορέσουν τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωζώνης ε, να πάρουν στα χέρια τους αυτή την πολιτική, πρέπει να περάσουμε από όλα τα κανάλια που φτάνουν προς αυτούς, με όλες τις γλώσσες που είναι κατανοητές ε, προς αυτούς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησα από όλους τους συνεργάτες μου να σταματήσουν να χρησιμοποιούν συντομογραφίες γιατί ε, χρησιμοποιώντας τα αρχικά οργανισμών απομονώνουν ε, τους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα που μιλάμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε μέσω τη γλώσσα μας να απευθυνθούμε προς πολίτες, προς καταναλωτές που δεν είναι εμπειρογνώμονες ε, σε θέματα νομισματικής πολιτικής, να καταλάβουν τι είναι η ΕΚΤ, σε τι χρησιμεύει, ε, γιατί αποτελεί ένα στοιχείο περιφερειακής κυριαρχίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλα αυτά είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν και πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα θελήσει με τα χαράς να προχωρήσει σε μια διαφορετική προσέγγιση και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Okay, now the last speaker, uh, last... Τελευταία ερώτηση. Κούσμαν. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Εδώ είμαι δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει δίμηνο. Καλά να μιλήσω αγγλικά τότε. Should respect limit for, for interpreters. Uh, I agree with uh, many of my... Συμφωνώ με πολλούς από τους συναδέρφους που είπαν ότι η μη συμβατική νομισματική πολιτική ήταν αναγκαία για να αποφευθεί η κατάρρευση της Ευρωζώνης. Και συμφωνώ επίσης ότι η μη συμβατική νομισματική πολιτική ελοχεύει και κινδύνους. Θέλω λοιπόν να βασιστώ στην εμπειρία της δικιάς μου χώρας που είχαμε ένα πακέτο λιτότητας ε, με νομισματική παρέμβαση στην Πορτογαλία που οδήγησε σε πολύ μεγάλη ύφεση αλλά επιπλέον και σε μεγάλη αύξηση του χρέους αυτά τα χρόνια της λιτότητας. Τα προηγούμενα χρόνια η νέα πολιτική πλειοψηφία αντέστρεψε τα μέτρα και έτσι είχαμε τα καλύτερα χρόνια σε ανάπτυξη όσον αφορά τα χρόνια που είμαστε εμείς στο ευρώ, αλλά και την μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους. Οπότε, η συζήτηση που πρέπει να γίνει και αυτή είναι και ερώτηση που σας μεταφέρω είναι το εξής. Πιστεύετε ότι αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους της ε, ε, πολιτικής ε, μη συμβατικών μέτρων μήπως ε, οδηγεί σε ένα νέο προβληματισμό ή πιστεύετε ότι η σταθερότητα της Ευρωζώνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νομισματική πολιτική που συνδυάζεται με πολιτικές λιτότητας όπως είχαμε μέχρι τώρα. Μπορεί είναι καλύτερα δηλαδή να έχουμε κάποιο μείγμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να χαιρετήσω τις προσπάθειες της Πορτογαλίας και των το γάλλον που πέρασαν από μια τόσο δύσκολη περίοδο. Και δεν με εκπλήσει το ότι ε, η αναλογία ΑΕΠ χρέους βελτιώθηκε πάρα πολύ, γιατί άρχισε να αναπτύσσεται η Πορτογαλία βγαίνοντας από το πρόγραμμα. Και οι συνάδελφοι στο Δούνο του λένε ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, παρόλο που βέβαια για τρία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και χρειάστηκε να γίνουν πολλέ μεταρρυθμίσει. Πάντως και συμβαίνει συχνά όταν έχουμε πολιτικέ αλλαγέ. Οι επόμενοι ακολουθούν μετά από το σημείο δηλαδή που σταμάτησαν οι προηγούμενοι και εκείνοι υποφελούνται από τα θετικά αποτελέσματα. Πάντως ήταν πολύ θετικές οι εξελίξεις. Πάντως, διαφωνώ μαζί σας για το ότι οτιδήποτε εξωτερική τριγμή για την Ευρωζώνη ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να χρησιμοποιεί το μείγμα που λέτε. Σίγουρα χρειάζονται και μεταρρυθμίσεις που είτε ήδη γίνονται ή πρέπει να γίνουν περισσότερες. Πιστεύω δηλαδή τελικά ότι αυτά πρέπει να πηγαίνουν μαζί και με αυτό θα τελειώσω και δεν θέλω να σας επιβάλλω επιπλέον δύο λεπτά. Η συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της Ευρωζώνης, βάζοντας στο κέντρο τον άνθρωπο, είναι ε, αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και αυτό θα κάνω και εγώ ως επικεφαλής της ΕΚΤ. Είμαι έτοιμη να το κάνω και όσο μπορώ περισσότερο θα ενώσω δυνάμεις